Buonasera. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Άρχεται η συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας, γιατί είναι πολύ φορτωμένη και η σημερινή και η αυριανή μας ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε ανεφάλης χρονοτριβής. Θέλω να σα ενημερώσω ότι διάφορα μέλη της Επιτροπής μου μίλησαν για το να θέσουμε ένα προφορικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο ανακοίνωσης για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού 2009-2010. Αυτό το πρώτο έγγραφο, το οποίο δεν έχει εγκριθεί, έχει όμως την υπογραφή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Μπαρόζο, και προκάλεσε πολλές ανησυχίες. Θα ήθελα να σα ενημερώσω προς το παρόν ότι αύριο το πρωί στι 9 μαζί με τους συντονιστέ θα λάβουμε την απόφαση εάν θα υποβάλουμε ή όχι προφορικό ερώτημα για το θέμα αυτό. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει υιοθετηθεί από το σώμα των επιτρόπων. Αύριο εξάλλου το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια αντίδραση της Επιτρόπου Fisher η οποία δεν έχει εκφραστεί επί του κειμένου ακόμα. Όμως οι επιπτώσεις των προτάσεων δημιουργούν ανησυχίες. Και αύριο μαζί με τους συντονιστές θα προσμετρήσουμε αυτές τις αντιδράσεις για να δούμε αν τελικά θα υποβάλουμε την ε, προφορική ερώτηση ή όχι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα ξεκινάμε πάντως συνεδρία τη ε, δική μα επιτροπή. Πλέον υπό την αιγίδα της ε, Συνθήκης Λισαβόνας, η οποία θα τεθεί και επίσημα σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου. Χαίρομαι λοιπόν που ξεκινάμε τη σημερινή συνεδρίαση τονίζοντας τη σημασία για τη γεωργία και τη γεωργική ανάπτυξη της ε, θέσης σε ισχύ αυτής της συνθήκη. Το έχουμε πει πολλάκις και είναι προφανές ότι μαζί με τη σημασία του τομέα για τον οποίο εμείς ενδιαφερόμαστε, της Γεωργίας, θα πρέπει να αναλάβουμε όλη την ευθύνη που η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει σε αυτήν την Επιτροπή. Ε, θα είναι πολύ πιο σημαντικές από εδώ και στο εξής οι προτάσεις μας, οι παρεμβάσεις μας, μια και από την 1η Δεκεμβρίου και εφ' η Επιτροπή θα, αυτή εδώ η Επιτροπή θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Συμβούλιο Υπουργών. Γι' αυτό έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία, θα παίξουμε μεγαλύτερο ρόλο, θα κάνουμε περισσότερες προτάσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Εγκρίνουμε λοιπόν τώρα τα πρακτικά. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι τα πρακτικά της συνεδρίας της 12 Οκτωβρίου, 29 και 30 Σεπτεμβρίου ε, είναι, έχουν εγκριθεί. Πολύ ωραία. Σας ενημερώνω ότι περνάμε απευθείας στο web streaming. Έχουμε τη μετάφραση σε όλες τις ε, γλώσσες και ευχαριστώ τους διερμηνείς. Σημείο 4. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Γαλακτοπαραγωγών, την ΕΝΤΑ. Πρόκειται για μια οργάνωση που ασχολείται με τα συμφέροντα των παραγωγών, ε, έρχεται σε επαφή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με τον Κόντεξ Αλιμεντάριους και τον ΠΟΕ, δηλαδή διεθνείς οργανώσεις. Αυτή η οργάνωση ασχολείται με θέματα διατροφής, υγείας, ασφάλειας των τροφίμων, ε, βιωσιμότητας, διαχείρισης αγοράς κτλ. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Βέρνερ Μποκ, που είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής αυτής οργάνωσης Γαλακτοπαραγωγών που θα μας παρουσιάσει την άποψη της οργάνωσής του για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του γάλακτος. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις ιδέες του για την πιθανή λύση απέναντι στο πρόβλημα της αστάθειας των τιμών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόκ έχει το λόγο. Mr. Chairman. Yes, thank you very much. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Γαλακτοπαραγωγών για να σας παρουσιάσουμε τις προοπτικές ε, του κλάδου. Όπως είπατε, Πρόεδρε, η Ένωσή μας, η EDA, είναι μια οργάνωση μέτρα της Βρυξέλλες που εκπροσωπεί την ε, μεταπητική βιομηχανία στον τομέα του γάλακτος των ευρωπαϊκών ε, κρατών μελών προς τις ευρωπαϊκές αρχές και η βιομηχανία αυτή έχει κύκλο εργασιών περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία περίπου 400.000 εργαζομένων και πιο πολύ το άνω του 100% του γάλακτος που μεταποιείται στην Ευρώπη μετατρέπεται σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα από εταιρείε που εκπροσωπεί η EDA. Ο γαλακτοκομικός τομέας δεν είναι μόνο ένας τομέας ε, τροφίμων. Επί σειρά ε, επί πολλούς αιώνες συμβάλλει στην ε, σωστή και υγιεινή διατροφή των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ ο κλάδος επίσης συμβάλλει σημαντικά στην ε, κοινωνική και οικονομική δομή, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Πρόεδρε, στην έκθεση για την κατάσταση στην αγορά των γαλακτοκομικών το 2009 που παρουσιάστηκε στις 22 Ιουλίου φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο γαλακτοκομικός τομέας έχει δραματική, σημειώσει δραματική ε, επιδείνωση από το καλοκαίρι του 2008. Στα τρία τελευταία χρόνια όντως έχουμε δει ε, εξελίξεις στον κλάδο μας που δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ πριν. Καταρχάς το 2007 και 2008 μια έντονη αύξηση των τιμών σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά ε, τα δευτερεύοντα προϊόντα, όπως το βούτυρο, το αποβουτρωμένο σκόνη γάλακτος και το καθεξής. Αυτό ε, σήμαινε αύξηση των τιμών μέχρι 45 λεπτά ανά λίτρο και στη συνέχεια το 2008-2009 οι τιμές έπεσαν περίπου στα 20 έως 25 λεπτά ανά λίτρο και πέραν αυτών βλέπουμε ότι σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παραγωγή γάλακτος ε, έχει πέσει κάτω από τις ποσοστώσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξέλιξεις σε αυτές, Πρόεδρε, έχουν, ε, έχουν αποτελέσει το έναυσμα για πολλές συζητήσεις για το τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και ο γυναιμικός έλεγχος έχουν εισάγει αλλαγές στο περιβάλλον λειτουργίας του κλάδου μας. Η απόφαση για τις αλλαγές αυτές βασίστηκε και στις εσωτερικές ε, εσωτερικού παράγοντε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε παράγοντες που σχετίζονται με τι εξελίξει στο παγκόσμιο εμπόριο. Και όλα τα μέτρα μεταρρύθμισης ε, σκοπό είχαν να υπάρχει μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά για την παραγωγή, για την ε, οργάνωσή μας. Οι πρόσφατε εξελίξεις στην αγορά δεν αποτελούν λόγο για να αλλάξουμε την προσέγγιση μας ως προς την πολιτική όπως ορίζονται στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2003 και στον υγειονομικό έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί για τον γαλακτοκομικό κλάδο την πιο σημαντική αγορά στον κόσμο και από πλευρά γεωγραφικών όρων και από πλευρά κλιματολογικών όρων σε πολλές περιφέρειες οι συνθήκες είναι ευνοϊκές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκτενής γνώση για την, ε, γνώσεις για την ε, παραγωγή γάλακτος και την επεξεργασία και τη μεταποίηση του γάλακτος ε, ξεχωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα, ξεχωρίζουν, θα ξεχωρίζουν και στο μέλλον. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου των γαλακτοκομικών στην Ευρώπη είναι η μεγάλη ποικιλία δομών σε όλη την γαλακτοκομική αλυσίδα. Οι λιανικοί έμποροι μπορεί να αποτελούν τη βασική οδό παροχή των προϊόντων προς τον καταναλωτή, αλλά τα γαλακτοκομικά προϊόντα περνούν και από εναλλακτικέ οδούς, όπως το catering για παράδειγμα. Και υπάρχουν, ε, είναι μεγάλη η αγορά συστατικών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ε, και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από πλευράς προμήθειας έχουμε πολλές μεγάλες αλλά και μικρές φάρμες, φάρμες που ειδικεύονται στην παραγωγή γάλακτος, αλλά και ε, φάρμες οι οποίες παράγουν άλλα προϊόντα. Από πλευράς μεταποίησης έχουμε ε, παραγωγούς μεταποιητές για μεμονωμένα προϊόντα, αλλά και παραγωγούς μεταποιητές για μια ολοκληρή σειρά προϊόντων. Κάποιοι εξ αυτών ε, είναι σε περιφερειακό επίπεδο, άλλοι δραστηριοποιούνται σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Πολλά από τα προϊόντα είναι υψηλής αξίας, αλλά σημαντικά, σημαντικό τμήμα της αγοράς ε, εστιάζεται σε, σε προϊόντα ε, όπου ο ανταγωνισμός εστιάζεται στην ε, τιμή. Για παράδειγμα βούτυρο, υγρό γάλα, τυρί και ούτω καθεξής. Και κεντρική, κεντρικό ρόλο εδώ παίζει το, το φρέσκο γάλα, το μη επεξεργασμένο γάλα. Και πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο ότι στο σημείο αυτό ότι οι παραγωγοί και οι μεταπητές πολλές φορές δεν έχουν έλεγχο ούτε στο γάλα αλλά ούτε και στην διαδικασία και στις υπόλοιπες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Και επίσης να σημειώσουμε ότι στις φάρμες όπου ξεκινάει ουσιαστικά η προμήθεια στην βιομηχανία ξεκινάει πολλές φορές και η μεταποίηση. Για τον κλάδο λοιπόν αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει μία ενιαία λύση, μία ομοιόμορφη λύση για τις σχέσεις μεταξύ των ε, παραγόντων. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να νομοθετήσει για ένα, μια κοινή σύμβαση για όλο τον κλάδο, μια σύμβαση η οποία θα ήταν ε, συμβατή και κατάλληλη, αν θέλετε, με όλες, για όλες τις δομές εμπορικών ε, σχεδίων και σχέσεων. Δεν υπάρχει ένα ομοιόμορφο πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη όλους τους όρους που επηρεάζουν και τα ε, αγροκτήματα και τους μεταποιητές. Αν οι πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή πολιτική ε, στρεβλώσουν την αγορά φρέσκου γάλακτος, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα μπορέσουν οι μεταποιητές να ανακτήσουν αυτό το επιπλέον κόστος από τους ε, πελάτες τους οι μεταποιητές γάλακτος δεν θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμειχθεί στη διαδικασία καθορισμού των τιμών. Και οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση για την, τον καθορισμό των τιμών θα δημιουργήσει ανεπάρκειες και έτσι δεν θα ενταχθεί στο περιβάλλον αυτό της αγοράς. Με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για τον γαλακτοκομικό κλάδο η τάση σε ό,τι αφορά τις τιμές θα τεθεί από την αγορά προϊόντων. Είναι τόσο σημαντικά τα προϊόντα αυτά για τις τιμές, γιατί η δυνατότητα να περάσει το φρέσκο γάλα προς τις μεταπητικές βιομηχανίες είναι καθοριστική και αυτό είδαμε σε διάφορες χώρες το 2007 και το 2008. Ο, τότε οι τιμές των προϊόντων α, αυξάνονταν και οι αγρότες πέρασαν από την παροχή γάλακτος στις ε, πελάτες στους μεταποιητές. Και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας αποδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή αγορά για το φρέσκο γάλα λειτουργεί Ε, επαρκώς προκειμένου να έχουν οι αγρότες ε, σωστή τιμή για το γάλα. Η οργάνωσή μας, η ένωσή μας θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος για παρέμβαση. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε τη δυνατότητα ε, να χορηγήσουμε στους παράγοντες της αγοράς τα κατάλληλα εργαλεία για να παραμείνει η δράση τους επικερδής. Η Ένωση Καλακτοπαραγωγών Πρόεδρε ζήτησε από το Πανεπιστήμιο του Κόρκ να ε, διενεργήσει μια έρευνα για την ε, σταθερότητα ημίτων τιμών στον γαλακτοκοπικό κλάδο. Και η έρευνα αυτή παρουσιάστηκε σε ένα ετήσιο κογκρέσο της Ένωσής μας τον προηγούμενο μήνα στην Πρατισλάβα διατίθεται και στην ιστοσελίδα μας. Μέχρι το 2003 η αστάθεια των τιμών στον κλάδο ήταν πολύ χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα όμως με την κατάργηση της πολιτικής της γαλακτοκομικής αγοράς στα πλαίσια της ΚΑΠ θα αυξηθεί και πλέον θα καταστεί εγγενής ε, στοιχείο αυτή η αστάθεια των τιμών και στην ευρωπαϊκή αγορά. Ουσιαστικά η αστάθεια των τιμών σε μεγάλο βαθμό είναι κάτι το θεμητό προκειμένου να λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο η αγορά. Ωστόσο, η ακραία αστάθεια των τιμών είναι κάτι το ανεπιθύμητο, γιατί στρεβλώνει την αγορά. Η λειτουργία σε μια σταθή αγορά προϋποθέτει την χρήση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες ε, συμβάσεις μελλοντικής ισχύω και συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτά τα ιδιωτικά ουσιαστικά όργανα δεν θα μειώσουν την αστάθεια των τιμών, αλλά μπορεί να περιορίσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η αστάθεια των τιμών για τους φορείς. Μόνο τα δημόσια μέσα μπορούν να πραγματικά να μειώσουν την αστάθεια των τιμών. Η EDA λοιπόν ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα ενός συστήματος ενδεχομένω για την ε, παρέμβαση σε ένα επίπεδο, αν επίπεδο δικτύου ασφαλείας για την ε, διαχείριση των στρατηγικών αποθεμάτων για να περιορίσει τις ακραίες καταστάσεις στην αστάθεια των τιμών. για μια αποδοτική αγορά για τον γραφτοκομικό κλάδο, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν σταθερές πολιτικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την μεταρρύθμιση της, ε, του 2003 και με τον υγειονομικό έλεγχο ορίστηκαν σαφείς ε, γραμμές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσει αυτές τις γραμμές τώρα. Θεωρούμε ότι ο βασικός κίνδυνος σήμερα είναι οι διάφορες πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη που μπορεί να οδηγήσουν σε πανεθνικοποίηση των πολιτικών για τον γαλακτοκομικό κλάδο, όχι μόνο για τις παρεμβάσεις ε, στην αγορά, αλλά και οι βασικές, αν θέλετε, οι βασικές αλλαγές, οι βασικές διαφορές μεταξύ των χωρών θα περιορίσουν τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, για να προσανατολιστεί ο κλάδος πιο πολύ στην αγορά, χρειάζονται εργαλεία τα οποία θα επιτρέψουν στον κλάδο να λειτουργήσει όντω στην αγορά. Και γι' αυτό λοιπόν ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα ενσωματώνει όλε τι πρωτοβουλίε όλων των γενικών διευθύνσεων τη Επιτροπή. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων είναι πολύ σημαντική. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία για να υπάρξει ευαισθητοποίηση για την υψηλή ποιότητα προϊόντων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να δοθούν στους ε, καταναλωτές πιο πολλές πληροφορίες για τα πρότυπα ε, παραγωγής που πληρώνουν κάθε μέρα. Τα διαφορετικά πρότυπα που έχουμε είναι καλά προσαρμοσμένα στα συγκεκριμένα προϊόντα και διασφαλίζουν ένα ίσο, αν θέλετε, ίσους όρους ανταγωνισμού στην Ευρώπη και καλή φήμη μας στις εξαγωγές. Οποιαδήποτε αλλαγή προς την απλοποίηση θα πρέπει να κρατήσει αυτή την ευελιξία για τους διάφορους κλάδους. Και είμαστε πεπισμένοι ότι η ισχυρή βάση, αν θέλετε, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία διασφαλίζει την καλή επισκόπηση όλων των ενδεχόμενων ε, επιπτώσεων στον κλάδο. Πρόεδρε, μία άλλη λύση για να διευκολύνουμε τις αγορές είναι να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η υποχρεωτική επισήμανση της ε, χώρας προέλευσης ε, είναι έντονα αντίθετη με αυτή την, με αυτή την αρχή. οι πληροφορίες που δίνονται στον καταναλωτή με την αναγκαστική επισήμανση ουσιαστικά προκαλούν μεγαλύτερη σύγχυση παρά βοηθούν τον καταναλωτή σε ό,τι αφορά αυτή την απόφαση για την αγορά. Θεωρούμε ότι με τις γεωργικές ενδείξεις έχουμε καλύτερες ε, επισημάνσεις. Για παράδειγμα, έχουμε το PDA, το PGI, το TSG. Έχουμε τρεις επισημάνσεις υψηλής αξίας, τις οποίες θα πρέπει να προστατεύσουμε και να τις τονίσουμε. Και σε ό,τι αφορά τη διατροφή και τις ε, κανονισμούς για την ε, υγεία, για την επισήμανση και τις χρήσεις. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Συζητάτε τώρα, για παράδειγμα, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ρύθμιση για την ε, ενημέρωση σχετικά με τα διατροφικά προϊόντα προς τους καταναλωτές. Πέραν αυτών, καθώς ε, συνεχίζονται οι συζητήσεις για τα διάφορα ε, προφίλ, ε, διατροφικά προφίλ, θεωρούμε ότι αυτές, αυτοί οι κανονισμοί είναι σημαντικοί προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα των προϊόντων αυτών για τους καταναλωτές. Ευχαριστούμε Πρόεδρε, για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε να σας παρουσιάσουμε αυτά τα σημαντικά στοιχεία τα οποία συχνά ε, τονίζουμε στις παρουσιάσεις μας. Κύριε Μποκ, ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση. Ο κύριος Ράσμουσεν, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, είναι στην αίθουσα και μετά τη συζήτηση θα του δώσω το λόγο για να παρέμβει και εκείνος. Ε, Μαγκίνες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπρόκ, για την παρουσίασή σας. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα ε, σχόλιά σας για ε, το πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι η υπερβολική αστάθεια των ε, τιμών και για τους παραγωγούς και για τους μεταποιητές. Παρακαλώ, σχολιάστε μας ε, τι θα γίνει όταν καταργηθούν οι ποσοστώσεις το 2015 χωρίς πραγματικούς μηχανισμούς υποστήριξης αγοράς. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια ανησυχία για τι σχέδια έχει η Κομισιόν για να υποστηρίξει την αγορά ε, των γαλακτοκομικών όταν φύγουν οι ποσοστώσεις. Και για να γίνει αυτή η κατάργηση θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια σαφήνεια για τους μηχανισμούς που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσετε το εξή. Μιλάμε για τους αγρότες οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο προσανατολισμό τώρα προς την αγορά και ξεχνάμε ότι σχεδιάζουν την παραγωγή. Ίσως την τιμή που οι τιμές είναι ψηλά, αλλά το πραγματικό γάλα παράγεται μια χρονιά μετά. Ε, επομένως, ε, δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις υψηλές τιμές. Ε, συχνά η ε, υπερπαραγωγή, ας πούμε, τελικά τους γυρνάει μπούμεραγκ, γιατί έχουν φύγει οι παχές αγελάδες όταν παράγουν το γάλα. Επίσης μιλήσατε για τις συμβάσεις και ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ε, μπει στη μέση ανάμεσα στους παραγωγούς και τους μεταποιητές. Μιλάμε για ιδιωτικές συμβάσεις και τι σχέδια υπάρχουν για αυτά. Θα ήθελα να σχολιάσετε για το κατά πόσον ε, βελτιώνεται ο τομέας των γαλακτοκομικών χάρη σε αυτά τα συμβόλαια. Ποιες είναι οι απόψεις σας για αυτό το θέμα. Εγώ θα ανησυχούσα ε, για οποιασδήποτε έτσι, προσπάθειες για να απελευθερωθούν ε, αυτά τα συμβόλαια. Ε, ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις ε, απαντήσεις ε, του κύριου Μπόκ. Ο κύριος Σικέρσκι. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες, αν έχετε βέβαια, για το ποια είναι η μορφή ιδιοκτησίας των εταιριών που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γαλακτοπαραγωγών. Δηλαδή, τι είδου μορφή γεωργική ιδιοκτησία έχουμε. Είναι ιδιωτικέ ιδιωτικά τα αγροκτήματα, υπάρχουν συνεταιρισμοί γεωργικοί. Επίσης, ε, μιλήσατε για την κατάσταση στην ε, γεωργική μεταποίηση και τις ιδιαίτερες σχέσεις ε, που ισχύουν. Τι γίνεται μεταξύ των σχέσεων παραγωγών ε, των μεταποιητών αλλά και των λιανεμπόρων. Δηλαδή υπάρχουν ε, τρεις συνιστώσεις σε αυτό το τρίγωνο, ο παραγωγός, ο μεταποιητής και τα μεγάλα εμπορικά δίκτυα. Είπατε ότι είναι, ε, επειδή είναι διαιάζουσα η κατάσταση σε πολλές χώρες, δεν επιδέχεται ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση. Τότε Μήπως έπρεπε να ακούσουμε περισσότερο τη γνώμη των γεωργών. Γιατί φτάσαμε στην κατάσταση που φτάσαμε σήμερα. Ποια είναι η πρότασή σας για να εξασφαλιστεί μια σταθερότητα και της παραγωγής και των τιμών, για να μην υπάρχουν τέτοιες διακοιμάνσεις των τιμών. Τι είδους μηχανισμού ρύθμισης προτείνεται για να σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Και πώς βλέπετε το μέλλον, όπως ρώτησε η κυρία Μαγκίνες. Τι προοπτικές υπάρχουν. Είστε υπέρ των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, υπέρ της παράτασης και μετά το 2015. Και τι γίνεται με τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών εταιριών ε, και των, ε, της ευρωπαϊκής αγοράς σε σχέση με τις παγκόσμιες ε, αγορές, με την παγκόσμια αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άλτεντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσίαση που μας κάνατε. Δεν ε, μας είπατε κάτι ουσιαστικά πολύ καινούργια. Είναι διαπιστώσεις τις οποίες έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Αλλά σωστά επισημάνατε, και αυτό θα ήθελα να αναπτύξω, ότι, ότι δεν ε, επιθυμούμε να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών, αλλά θα ήθελα πιο πολλές πληροφορίες να μου δώσετε. Πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα σύστημα προκειμένου να αποφευθούν τέτοιες επερβολικές διακυμάνσεις. Γιατί πολλές φορές ακούω από διάφορους αγρότες, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ότι σκέφτονται να διαθέσουν την ε, παραγωγή γάλακτός τους σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ε, αν παραμένει τόσο χαμηλή η τιμή του γάλακτος και θα πρέπει να βρούμε ένα δίκτυο ασφαλείας προκειμένου να υπάρχουν δυνατότητες κρατικής παρέμβασης σε περιπτώσεις ε, εξαιρετικών διακυμάνσεων, αν θέλετε να απαντήσετε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Προέρχομαι από μια περιφέρεια όπου πάντα υποστηρίζονταν ο κλάδος με κρατικές ε, ενισχύσεις. Ε. Ωστόσο, πριν από κάποια χρόνια έκλεισε μια μεγάλη εγκατάσταση και εντό σύντομου χρονικού διαστήματος ε, τετραπλασιάστηκαν οι κρατικές επιδοτήσεις και αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε σκληρό τίμημα. Αν συμβεί το ίδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα είναι πολύ πιο τραγικέ οι επιπτώσει για τον καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα σύστημα το οποίο να προσανατολίζεται στην αγορά όντω και θα ήθελα η αγορά να βελτιώσει, αν θέλετε, να διορθώσει την όλη μα ε, ενέργεια. Αλλά ναι, σε περιπτώσεις ε, ακραίες θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης. Δεύτερη ερώτηση, πώς ε, θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα μπορεί να ε, αποβούν εις βάρος περιοχών που δεν έχουν σωστή παραγωγή, δεν είναι ανταγωνιστικές για την παραγωγή του γάλακτος. Και μία άλλη ερώτηση δραστηριοποιούμε σε μια περιφέρεια που υπάρχουν πολλοί παραγωγοί και μεγάλη παραγωγή. Μας καταπιέζει ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις η δύναμη της αγοράς. Και χρειαζόμαστε πολύ απλά οργάνωση και διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε σε σωστό επίπεδο. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το εμπόριο τα συνδικάτε ε, παίζουν ουσιαστικά με το εμπόριο, γιατί δεν μιλάμε για 30 μέρες, μιλάμε για 20 μέρες και αυτή την εβδομάδα παρευρέθηκα στο Παρίσι όπου και έμαθα ότι στη Γαλλία υπάρχει ένα ανάλογο σύστημα το οποίο ορίζεται κρατικά που μιλά για πληρωμή 21 ημερών. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μια ανάλογη ρύθμιση και για μας, να το σκεφτούμε από πολιτικής άποψης μετά. Από 30 ημέρες θα πρέπει για παράδειγμα ο κλάδος να πληρώνει υποχρεωτικά τους εργαζόμενους. Αυτό θα βελτίωνε δραστικά την κατάσταση και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να περάσουν ακριβώς τέτοιες ρυθμίσεις. Ευχαριστώ Albert. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καλεσμένο μας για το πώς επηρέασε το γαλακτοκομικό το, μάλλον οποια, οποιαδήποτε αλλαγή στο γαλακτοκομικό τομέα πώς θα επηρεάσει τον ΠΟΕ. Γιατί αν ε, αυξηθούν ε, οι τιμέ γάλακτος, προκειμένου να είναι κερδοφόρο ο, ο κλάδος, ο, οι γεωργοί θα, θα προσπαθήσουν να επεκταθούν, αλλά κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει ίσως διαταραχή στην παγκόσμια αγορά. Πώς πιστεύετε θα διδράσει ο ΠΟΕ σε μια τέτοια κατάσταση. Η κυρία Ντότ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα τη ρευστότητα ή της υπερβολικής μεταβλητότητας των τιμών. Στη Βόρεια Ιρλανδία αυτή η αστάθη των τιμών στο γαλακτοκομικό κλάδο επηρέασε αισθητά την ε, γενική οικονομία τη υπερβολικη μεταβλητοτητα Ιρλανδίας. Στη Βόρεια Ιρλανδία έχουμε ένα μικρό μόνο ποσοστό τη παραγωγή του ιρλανδιας στη βορεια ιρλανδια εχουμε ενα μικρο μονο ποσοστο τη παραγωγη του γαλακτο που διοχετεύεται στην αγορά. Το περισσότερο γάλα που παράγεται ε, ε, μετατρέπεται σε σκόνη. Οπότε η αστάθεια των τιμών είχε σημαντική επίπτωση και μετά το 2007 και μετά τη, με τη χρηματοπιστωτική κρίση πολλοί γεωργοί μας και κτηνοτρόφοι βρέθηκαν σε πολύ δινή οικονομική κατάσταση. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς της αγοράς και στις δύο πλευρές του φάσματος για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αστάθεια των τιμών του γάλακτος. Ο κλάδος στη Βόρεια Ιρλανδία μου λέει ότι μερικοί, αυξάνονται με, με, μερικοί ικανοποιούνται με την αύξηση των τιμών του γάλακτος, αλλά μπορεί αυτή η αύξηση των τιμών να οφείλεται στη χαμηλή παραγωγή ή στην α, ε, ε, έλλειψη της ε, προσφοράς. Μήπως όμως ε, μια μαζική ροή προϊόντων στην αγορά θα αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ε, προβεί σε περαιτέρω πρόταση να αναλύσει όλες τις επιπτώσεις της πρόσφατης αύξησης των τιμών προκειμένου ε, να μην διακυβευτεί το μέλλον της αγοράς στο βωμό ενός βραχυπρόθεσμου κέρδους. Uh, στο ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την επιρροή των σούπερ μάρκετ στις τιμές. Ο κύριος Γκάντφελπερ. γιατί ακόμη και αν μειώνονται οι τιμές ε, του γάλακτος για τους παραγωγούς, οι τιμές ε, στα σούπερ μάρκετ του γάλακτος δεν μειώνονται και επομένως δεν αποφελούνται οι καταναλωτές. Αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο για τους παραγωγούς του γάλακτος, αλλά και για τους μεταποιητές. Στην ε, παρουσίασή σας δεν μιλήσατε αναλυτικά για το θέμα αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας, τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Και εσείς πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ρωτάω αυτό γιατί στις διαπραγματεύσεις ε, ε, με τα σούπερ μάρκετ ε, εσείς και τα μέλη σας ουσιαστικά είσαστε συνομιλητής στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό σας ρωτάω λοιπόν εσάς αυτό το ερώτημα. Ο κύριος Μαρτίν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την παρουσίαση αυτή, μας είπατε ότι η αγορά είναι εντάξει, ότι δεν χρειαζόμαστε παρεμβάσεις, ότι όλοι έχουν σωστό εισόδημα, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι αν αυξηθεί η τιμή δύο λεπτά θα είναι σωστό το εισόδημα των αγροτών. Νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη δική σας, όχι των γεωργών. Μία συγκεκριμένη ερώτηση να κάνω. Αρνηθήκατε ότι την χρήση μ, γεωργικών ενδείξεων. Γιατί το απορρίπτεται αυτό ως μέτρο. Βλέπουμε ότι προς τα εκεί είναι η τάση και ότι ο καταναλωτής θέλει τα τοπικά προϊόντα. Και στη συνέχεια ανακύπτει το άλλο ερώτημα. Τι θα γίνει όταν εκπνεύσει η ρύθμιση τρέχουσα για τους ε, για τον γαλακτοκομικό κλάδο. Πώς φαντάζεστε ότι θα είναι οι καινούργιες ρυθμίσεις μετά τις ποσοστώσεις ουσιαστικά. Μία τελευταία ερώτηση. Το 7% εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο ισχύει ως ποσοστό ή έχουν μεταβληθεί τα αριθμητικά στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γαλακτοπαραγωγών για την παρουσίασή του που αντανακλά τη θέση του γαλακτοκομικού κλάδου. Εμάς μας ενδιαφέρουν όμως και άλλες απόψεις γιατί η δική του είναι αξιοσέβαστη αλλά είναι μεμονωμένη γιατί υπερασπίζεται τα αξιοσέβαστα δικαιώματα των μεταποιητών. Βέβαια, αυτή η συνεδρίαση και αυτή η κατάσταση λαμβάνει χώρα εν μέσω μια σημαντική χρηματοπιστωτική κρίση, όπου ένα σημαντικό τμήμα των Ευρωπαίων παραγωγών αντιμετωπίζουν τεράστιε δυσκολίε. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, το μοντέλο που είναι καλό για τη βιομηχανία, για τον κλάδο, δεν ε, είναι κατάλληλο για τους ε, γεωργούς, για τους παραγωγούς. Και ένα σύστημα μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα μόνο όταν ε, όλα τα τμήματα του συστήματος αντλούν κάποια ωφέλη από το σύστημα αυτό, από το μοντέλο αυτό. Ο κλάδος είναι υπέρ της, της τη της φιλελεύθερης λογικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που Δίχασε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγους μήνες όταν εξετάσαμε το check-up της Γεωργίας, το διαγνωστικό έλεγχο. Για το θέμα των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων δίχασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαιτία τη ε, διάσταση απόψεων που υπάρχουν μεταξύ τη μία πλευρά και τη άκρο νεοφιλελεύθερη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε είστε υπέρ επίση ενό μηχανισμού παρέμβαση και δικτύου δικλείδα ασφαλεία. Το θέμα είναι τι μηχανισμοί πρέπει να υιοθετηθούν για να αποφύγουμε τα δύο άκρα αυτή τη ρευστότητα των τιμών. Θα ήθελα όμω ε, κάποιε περισσότερε λεπτομέρειε. Τι είδου ε, δίκτυο ασφαλεία θέλετε. Το δίκτυο ασφαλεία δεν είναι μηχανισμό παρέμβαση. Είναι ένα επίπεδο που εμποδίζει ουσιαστικά του παραγωγού ε, να εξαφανιστούν τους βοηθάει απλώς να επιβιώνουν. Αυτό που συμβαίνει και η λύση αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Θα ήθελα λοιπόν περαιτέρω διευκρινήσεις. Ποιοι μηχανισμοί πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν σε αυτό το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο και μπορούν να υιοθετηθούν από τους πολιτικούς ηθήνοντες. Γιατί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει όλο και περισσότερο λόγο στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Τρεις ερωτήσεις έχω να απευθύνω. Πρώτη. Διαπίστωση, αν συμφωνείτε ρωτάω. Θεωρώ ότι η παραγωγή του γάλακτος στο μέλλον θα πρέπει να προσανατολιστεί πιο πολύ στην αγορά από ό,τι έως τώρα. Συμφωνείτε? Δεύτερη. Πολλοί συνάδελφοι το έθιξαν ε, παρομοίως τουλάχιστον. Βλέπουμε διακυμάνσεις τιμών έντονες τον τελευταίο καιρό και διακυμάνσεις στην αγορά. Πώς θα μπορούσαμε μέσω των σωστών συμβατικών σχέσεων να ρυθμίσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διακυμάνσεις έτοιμων Γιατί έχουμε το φαινόμενο το εξής, ε, τι γίνεται με τις συμβατικές σχέσεις, την υπερβολική παραγωγή, τη χαμηλή ζήτηση και ούτω καθεξής. Στη Γερμανία συζητιέται ένα σύστημα συμβατικό με διάφορα ύψη τιμών, με διαφορετική αποζημίωση, με διαφορετικό δηλαδή ποσό βάσης. Και τρίτη ερώτηση. Θεωρείτε, πώς θεωρείτε και πού θεωρείτε ότι στο μέλλον στο μέλλον, τονίζω, πού θα πρέπει να αναμειχθεί η πολιτική και πού όχι. Πού θεωρείτε ότι μπαίνει το όριο, να πείτε δηλαδή ότι κοιτάξτε εδώ εμείς θα διαμορφώσουμε την κατάσταση στην αγορά του γάλακτος, αλλά από το σημείο αυτό και πέρα χρειαζόμαστε βοήθεια από την πολιτική. Madame Kostinger. Kostinger. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Κύριε Μπόκ, είπατε ότι είναι πολύ ευνοϊκή η κατάσταση στην Ευρώπη ε, για την αγορά γάλακτος, αλλά υπάρχουν και μειονεκτούσες περιοχές, όπως για παράδειγμα οι ορεινές, όπου παρόλα αυτά ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εκεί πολλές θέσεις εργασίας. πώς θεωρείτε ότι στο μέλλον ε, θα μπορούμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα των περιοχών αυτών και όπως είπατε και στην παρουσίασή σας, δεν εξαντλείται η ποσόστοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε επιδιώξει σε, αυτό το επίπεδο για να προσθεθούν, για παράδειγμα, στην αγορά νέα κοινοτομικά προϊόντα. Grazie, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια στοιχεία που προκύπτουν από ένα έγγραφο της ε, Επιτροπής Βιομηχανίας που σε ένα κεφάλαιο για τον αγροπιστιστικό κλάδο λέει ότι σύσσωμος ο κλάδος, αναφέρεται στη σελίδα 4 του εγγράφου, ότι το πραγματικό, το ουσιαστικό πρόβλημα σήμερα για τον κλάδο αυτό είναι το, κόστος, το, το υψηλό κόστος της πρώτης ύλη. Δεν μπορεί ο κλάδος να είναι ανταγωνιστικός με τόσο υψηλό, υψηλές, ακριβές πρώτες για να είναι ανταγωνιστικός στην παγκόσμια αγορά. Ε, φαίνεται ότι και το 2009 η τιμή των πρώτων υλών είναι υψηλή. Αυτό πιστεύει ο αγοραπιστωστικός κλάδος. Επίσης, στον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου του 2009 της Danone, που είναι μεγάλη γαλακτοκομική βιομηχανία, αναφέρεται ρητά ότι το κέρδος της επιχείρησης αυτής της Danone για το πρώτο εξάμεινο οφείλεται στις τιμές γάλακτος που ήταν ε, πιο χαμηλές από ποτέ και χάρη σε αυτές τις χαμηλές τιμές στο γάλακτος αύξησε η Danone τα κέρδη της. Φαίνεται ότι υπάρχει μια απόλυτη αντίφαση μεταξύ των δύο δηλώσεων, γιατί αφενό ο αγορεπιστικό κλάδο που θέλει χαμηλέ τιμέ παραπονιέται για την ακρίβεια των τιμών, αφετέρου έχουμε του ε, γεωργούς που δεν μπορούν καν να καλύψουν ε, τις δαπάνες τους, τα έξοδα της ε, εκμετάλλευσής τους και βγαίνουν στους δρόμους. Θα στερηθούμε το γάλα στην Ευρώπη αν δεν επιτρέψουμε στους παραγωγούς, τους γεωργούς να καλύπτουν τα, τις δαπάνες τους, τουλάχιστον τα έξοδά τους και έχουν τόσο χαμηλό κόστος ε, τιμών. Είστε υπέρ κάποιων μηχανισμών ελέγχου της παραγωγής προκειμένου να υπάρξει μια συνάφεια μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, γιατί η σχέση προσφοράς και ζήτησης καθορίζει την τιμή. Δεύτερον, συμφωνείτε με κάποιες ε, διαπαγγελματικές συμφωνίες μεταξύ ε, παραγωγών και βιομηχάνων να καθοριστούν κάποιες ε, τιμές γάλακτος όπου η βασική τιμή θα είναι υποχρεωτική και με βάση κάποιο κόστος παραγωγής που θα επιτρέπει στους ε, γεωργούς να επιβιώσουν. Και κάτι άσχετο με το γάλα γαλαγελάδος, είχαμε μια συζήτηση πριν αρχίσει η συνεδρίαση και αφορά μέσα και το θέμα αυτό ο κλάδος της παραγωγής ε, πρόβιο γάλατος και αυτός διανύει κρίση, ειδικά στη Γαλλία και την Ιταλία, για πολύ διαφορετικούς όμως λόγους. Σήμερα η παραγωγή πρόβιο γάλακτος αντιμετωπίζουν αντίστοιχη κατάσταση με αυτή των ε, παραγωγών γάλακτος αγελάδος. Θα ήθελα λοιπόν ε, και σας απευθύνω έκκληση γι' αυτό να ζητήσουμε για να βοηθήσουμε και αυτό το σημαντικό κλάδο και μάλιστα σε δύσκολες, σε δύσκολες περιοχές της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Γαλλίας να εφαρμόσουμε και για το πρόβιο γάλα αντίστοιχα μέτρα με αυτά που εφαρμόσαμε για το γελαδινό γάλα για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να εξέλθουν από την κρίση. Συναφές πρόβλημα, αλλά και ο κλάδος του, των παραγωγών πρόβιο γάλακτος αντιμετωπίζει κρίση. Σμίτ, έχει το λόγο. Thank you, President. I uh, will... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο, γιατί δεν θέλω να επαναλάβω κάποια πράγματα που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Με ενδιαφέρει το ερώτημα και η απάντηση στο ερώτημα της κυρίας Μαγκίνης Νομίζω ότι είναι ουσιαστικό για την, τις επιπτώσεις της πολιτικής που θέλουμε να προωθήσουμε. Ένα συγκεκριμένο σημείο. Ε, την εχθρότητα της ε, ε, ΕΝΤΑ για την υποχρεωτική επισήμανση και την ανείχνευση της προέλευσης. Αυτό μου φαίνεται περίεργο. η παραγωγή στην Σκοτία θέλουν τέτοια υποχρεωτική επισήμανση. Ε, νομίζω ότι αυτό θέλουν οι καταναλωτέ ε, να ξέρουν. Και το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ε, η ποιότητα, η στρατηγική ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για να εξασφαλιστεί η ποιότητα. Θα ήθελα να μου πείτε, εσεί μιλάτε φυσικά για τα συμφέροντα τη δική σας οργάνωση και θέλετε να παράγετε, ας πούμε, ένα γεωργικό προϊόν, όχι ένα απλό προϊόν αλλά θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε, να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κυρία Μετάλβες. Ο κύριος. Ευχαριστούμε κύριε Μπακ. Ο κύριος Μπακ επέμεινε ιδιαίτερα στην παρουσίασή του στην ε, ρευστότητα των τιμών. Αλλά δεν μας περιέγραψε κάποια πολύ καθοριστικά χαρακτηριστικά, που είναι οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν στην αναλογή της ε, κατανομής των εισοδημάτων στη γαλακτοκομική αλυσίδα, γιατί η τιμή της πρώτης ύλης αυξήθηκε, η τιμή της παραγωγής επίσης αυξήθηκε και οι τιμές ε, των προϊόντων πληρώνει ο καταναλωτής. Αλλά κάποια αργότερα έπεσαν οι τιμές πρώτη ύλες και έπεσε και η τιμή παραγωγής, αλλά η τιμή του τελικού προϊόντος παρέμεινε υψηλή. Οπότε διαταράχθηκε ε, η σχέση, η αρχική σχέση μεταξύ του κέρδους που αποκόμισαν οι παραγωγοί και του κέρδους που αποκόμισαν οι, οι λιανέμποροι. Ποια είναι η γνώμη σας ε, για τον τρόπο που λειτουργήσε η αγορά ε, και πώς ε, λειτουργεί η αγορά μεταξύ των παραγωγών και των μεταποιητών και της τελικής αλυσίδα ε, εμπορίου. Γιατί θα πρέπει να αποκατασταθεί μια τέτοια ισορροπία. Γιατί είναι σημαντική η ρύθμιση και είναι σημαντική και η συμφωνία με την άλλη πλευρά, δηλαδή με τους παραγωγούς γάλακτος όχι μόνο με τους βιομηχάνους ή με τους μεταπίτες. Έτσι εφαρμόζουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη σε όλη τη διάρκεια της αλυσίδας ε, γαλακτοπαραγωγής, κάτι που είσαι στο δικό σας μοντέλο δεν το λάβατε υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ολένιτσακ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Έχω μερικές ερωτήσεις και δύο παρατηρήσεις. Θα ήθελα καταρχήν να μιλήσουμε ευρύτερα για την κρίση στον τομέα. Όχι μόνο για τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις και για την αγορά, αλλά μιλήσουμε, να μιλήσουμε και για τις επενδύσεις που έγιναν από το γαλακτοκομικό κλάδο τα τελευταία χρόνια. Γιατί χάρη σε επενδύσεις αυτές εξυγχρονίστηκε ο κλάδος και έγινε πιο ανταγωνιστικός στην παγκόσμια αγορά. Έχω και μία σχετική ερώτηση προς τον κύριο Μπακ. Πώς εκτιμάτε το ύψος αυτών των επενδύσεων και έγιναν, είχαν πραγματικά αντίκτυπο, δηλαδή επέδρασαν θετικά στη βελτίωση του κλάδου. Πώς επηρέασαν τις συνθήκες και τη λειτουργία της γεωργίας. Γιατί όταν είχαμε την καλύτερη συγκυρία ε, στην γαλακτοκομική παραγωγή, τότε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης επένδυσαν τεράστια κονδύλια στην διεύρυνση της παραγωγής, στην αύξηση της παραγωγής και ίσως σε κάποιο βαθμό και αυτή η επέκταση μπορεί να συνέβαλε στην σημερινή κρίση. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση, ποιος είναι ο δικός σας απολογισμός. Έγιναν κάποιες μελέτες για το τι βοήθεια θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια ο κλάδος. Και δεν μιλάω μόνο για την παραγωγή και τις εξαγωγές. Και ως προς τις επενδύσεις τι ενίσχυση θα χρειαστεί ο κλάδος. Γιατί πολλές φορές και οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται με κοινοτική συμμετοχή ή τουλάχιστον με κοινοτική συγχρηματοδότηση. Τρίτη και τελευταία ερώτηση σε σχέση με αυτά που είπαν ο κύριος Μποβέ και ο κύριος Σεκέρσκι. Το 2008 που ήταν το απόγειο της κρίσης, τι έγινε με τις εταιρείες και ποια είναι τα σχέδια για το 2007, γιατί πολλές επιχειρήσεις δήλωσαν κέρδη. Τα μερίσματα πού θα κατανεμηθούν, θα αφιερωθούν στις επενδύσεις αυτού του κλάδου. Πώς θα παρέμβουμε στην αγορά. Σε ποιο θα φτάσει αυτό το κέρδος που δήλωσαν πολλές επιχειρήσεις παραγωγής γάλακτος. Ευχαριστώ. Oui. Merci, Monsieur le Président. Deux... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερώτησεις. Η γαλακτοκομική παραγωγή ε, είναι συνήθως, ε, έχει συνήθως χαμηλές τιμές ε, στην επικρατεία μας. Γι' αυτό έχει νόημα να έχουμε ε, μια δημόσια πολιτική και να συγκεντρώσουμε την παραγωγή σε περιοχές όπου το κόστος συλλογής του γάλακτος δεν είναι τόσο σημαντικό. Τι περιμένετε από την κοινότητα ούτως ώστε να αντιστοιχίσει τους δύο, τα δύο σκέλη της ε, εξίσωση. Επίση, σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η σκόνη γάλακτος ε, ήταν ο ρυθμιστικός παράγοντας ε, της τιμής του γάλακτο. Η βιομηχανία σας επενδύει σήμερα στην έρευνα και στην μη επισητιστική χρήση των πλεονασμάτων γάλακτος και σκόνη γάλακτος που φτάνει σε, που φτάνει εσάς δυνάμει των συμβάσεων που έχετε με τους παραγωγούς. Κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στη Σοβιετική Ένωση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε την ε, τιμή παραγωγής και την ε, τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής από τις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι με αυτή την αρχή. Διαπιστώνω ότι τουλάχιστον στη χώρα μου, εκεί όπου υπάρχει συνεταιρισμός των παραγωγών και όπου έχει δύναμη, μιλάω για το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου, η παραγωγή που δίνουν το γάλα τους σε, αυτή την, σε αυτό το συνεταιρισμό ε, πληρώνονται καλύτερα από εκείνους που δίνουν το γάλα τους σε μια γαλακτοκομική εταιρεία, ας πούμε, στη Γερμανία. Ε, αυτοί ε, θεωρούσαν ότι θα τους έδιναν οι Γερμανοί καλύτερες τιμές, γι' αυτό έφυγαν από το συνεταιρισμό. Ε, παραλίγο να σκοτώσουν μάλιστα, να τον υπο, υποσκάψουν τον συνεταιρισμό Πιστεύοντα λοιπόν ότι θα έχουν καλύτερε τιμέ, αλλά νομίζω ότι τώρα ε, πάει καλά ο συνεταιρισμό. Φυσικά η παραγωγή είναι ελεύθερη να ενταχθούν σε, μια, σε ένα συνεταιρισμό ή όχι, αλλά νομίζω ότι θα είναι πιο δυνατή ως ε, εταίρο στην αγορά αν το κάνουν, μέσω ενό συνεταιρισμού λοιπόν. Ε, σε αυτή την συνεχιζόμενη κρίση νομίζω θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα της αγοράς, όλα τα εργαλεία της αγοράς που ευτυχώς ε, διατηρήσαμε. Η κυρία Φίσορ Μπόιλ ήθελε να τα καταργήσει όλα αυτά τα μέσα, την ρυθμίση της αγοράς, την παρέμβαση, τις επιστροφές, όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ε, σωστά και με σύνεση μέσα στη σημερινή κρίση. Ε, πρόσφατα ε, αυξάνονται οι τιμές, ευτυχώ, ε, αυξήθηκαν οι τιμές ευτυχώς. Σε αυτή τη φάση λοιπόν θα πρέπει η Κομισιόν να μην πουλήσει τώρα τα αποθέματα, να μην τα αδιοχετεύσει στην αγορά. Γιατί θα πρέπει να περιμένει λιγάκι για να μην προκαλέσει εκ νέου πρόβλημα και να μην δημιουργήσει κρίση στις τιμές. Νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουμε τα εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα που έχουν ληφθεί για να επιτρέψουν ε, βραχυπρόθεσμα στους παραγωγούς να διανύσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. σε διάφορες χώρες έχουμε τέτοια μέτρα και στη δική μου χώρα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ σωστά και με σύνεση τα 280 δισεκατομμύρια του Γαλακτοκομικού Ταμείου για να αντιμετωπίσουμε τα, τα προβλήματα. Βέβαια, είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτά τα δισεκατομμύρια, αλλά ε, καλύτερα μια σταγόνα παρά τίποτα. Ίσως η Κομισιόν, αν ξαναψάξει εκεί στο βάθος των συρταριών της, θα μπορούσε να βρει και κάποια άλλα μέσα και κάποια άλλα κονδύλια. Θυμάμαι ότι όταν σώσαμε το Γαλιλαίο, το κάναμε με τα πλεονάσματα του γεωργικού προϋπολογισμού. Θα μπορούσαμε ίσως αυτή τη δύσκολη κατάσταση να δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε τίποτα υπόλοιπα παραδείγματο χάρη 500-600 εκατομμύρια, αυτά που ζητήσαμε. Τώρα, για τις ποσοστώσει, δυστυχώ η ίδια η παραγωγή είναι διαιρεμένη. Πρέπει να τις κρατήσουμε ή πρέπει να τις καταργήσουμε. Ε, αν συμφωνούσαν, εγώ θα ήθελα να τους βοηθήσουμε να συμφωνήσουν. Γιατί, διαρωτώ με, μήπως είναι παράλογο να καταργήσουμε τις ποσοστώσεις στη σημερινή συγκυρία. Ξέρω ότι λήφθηκε απόφαση, αλλά μπορούμε πάντα να αλλάξουμε μια απόφαση, η οποία λήφθηκε σε μια χρονική στιγμή όπου η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική από τη σημερινή. Αν υπήρχε μια πλειοψηφία παραγωγών που ζητούσαν τη διατήρηση των ποσοστώσεων πέρα από το 2015, νομίζω ότι θα το θεωρούσα ικανοποιητικό για αυτή την ε, κατάσταση και θα το δεχόμουν. Γιατί δεν ξέρουμε πώς αυτή η κατάργηση θα επηρεάσει τη διατήρηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε ένα επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλούς λόγους. Και σε όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να διατηρήσουμε ένα ελάχιστο αριθμό τέτοιων εκμεταλλεύσεων. Η απουσία κοινή γεωργική πολιτική θα μα κοστίσει πολύ πιο ακριβά. Πολύ πιο ακριβά θα κοστίσει στην ε, κοινωνία μα. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Γιατί οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απουσία ενός κατάλληλου ιστού στην Ήπεθρο, ε, ενός κατάλληλου αριθμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλες τις περιοχές, θα μας κοστίσει πανάκριβα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να ξανασκεφτούμε μήπως πρέπει να λάβουμε τέτοιου τύπου μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα κλείνουμε τον κατάλογο των ομιλητών με την κυρία Σαλντεμός. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά θα ήθελα πρώτα να πω ότι αν μη τι άλλο σε κάτι συμφωνώ με την κυρία Λούλινγκ. Γιατί το να πιστεύει κανεί ότι οι Βρυξέλλε μπορεί να αποφασίζουν για την τιμή των γαλακτοκομικών προϊόντων και αυτό θα δώσει μια θαυματουργή λύση, διαφωνώ. Αυτό θα πρέπει να ευνοήσει και του παραγωγού. Γιατί κανένα δεν μίλησε για του καταναλωτέ. Αν οι τιμέ καθοριστούν στι Βρυξέλλες, αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, θα πληρώνουν δύο φορέ ε, την τιμή του γάλακτος μία φορά χρηματοδοτώντας την ενίσχυση προς τον παραγωγό και τη δεύτερη φορά πληρώνοντας ακριβά το γάλα στα καταστήματα, στα εμπορικά καταστήματα και στο σούπερ μάρκετ. Τι θα κάνετε λοιπόν για να αυξήσετε τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των τιμών. Γιατί διανύουμε μια οικονομική κρίση και η τιμή του γάλακτος είναι υψηλή για τους καταναλωτές σήμερα. Η τελική τιμή του γάλακτος είναι ακριβή. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μία λύση. Τι μπορείτε εσείς να κάνετε για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια απέναντι στους καταναλωτές, γιατί ο τρόπος καθορισμού των τιμών είναι ύποπτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Σα ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Πολλέ ερωτήσει ακούσαμε. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το εξή. Οι επιχειρήσει τη EDA είναι ικανοποιημένε με την δομή που έχουν. Ποια είναι η δομή που θεωρείτε ότι είναι βέλτιστη και πώ θεωρείτε ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί συγκεκριμένα η στρατηγική σα για το μέλλον. Ε, ο καθένα θα ακολουθήσει τον δρόμο του ή έχετε μια κοινή γραμμή. Κύριε Μπόκ, ακούσατε πολλοί άριθμες ε, ερωτήσεις, ε, προβληματισμούς. Ε, φαντάζομαι ότι μερικές είναι εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της οργάνωσης που εκπροσωπείτε. Περιμένουμε πάντως την απάντησή σας και συνεχεία θα δώσω το λόγο στον κύριο Ράσμουσεν για να παρουσιάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις που μου θέσατε όσο μπορώ. Και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων εάν αφήσω εκτός κάποιες ερωτήσεις, αν έχω ξεχάσει κάποιες ερωτήσεις, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλές. Καταρχάς, θα ήθελα να σας εξηγήσω τι κάναμε το 2003 με το health check. Γιατί αυτή την πραγματικότητα βιώνουμε σήμερα με το διαγνωστικό έλεγχο. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, μείωσε κατά 15 με 25% τις τιμές παρέμβασης. Και αυτή η μείωση των τιμών της παρέμβασης αντισταθμίστηκε με κάποια συμπριμοδοτήσεις για τους ε, γαλακτοπαραγωγούς 3,5 ε, λεπτά το λίτρο. Το σύστημα των ποσοστώσεων θα σταματήσει το 2015 και δεν υπάρχει πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρατείνει τις ποσοστώσεις. Και στη συμφωνία για το διαγνωστικό έλεγχο όλοι συμφωνήσαμε ότι θα υπάρχει μια βαθμία αύξηση της παραγωγής, ούτω ώστε να προσγειωθούμε ομαλά και όχι ανώμαλα. Αυτές είναι οι πραγματικότητες που αντιμετωπίζουμε σήμερα και εμείς ως οργάνωση των γαλακτοπαραγωγών συμφωνήσαμε με όλες αυτές τις αποφάσεις. Συμφώνησε η EDA, η οργάνωσή μας. Τώρα, πιο μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά τις προοπτικές των αγορών και ποιες είναι οι προοπτικές μακροπρόθεσμα. Όλες οι εκθέσεις δείχνουν ότι μακροπρόθεσμα η ζήτηση θα αυξηθεί περισσότερο από την παραγωγή σε όλο τον κόσμο. ειδικά στις μη αναπτυσσόμενες χώρες. Συνολικά λοιπόν, παγκόσμια, η κατάσταση δεν θα είναι άσχημη. Τώρα, για την, τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Το 8 με 10% ε, ετησίως εξάγεται σε τρίτες χώρες. Τώρα, τι γίνεται παγκόσμια, τι, τι μπαίνει στο εμπόριο παγκόσμια. Είναι το 4 με 5 της παγκόσμιας παραγωγής που γίνεται αντικείμενο μέσω συμβολέων. Παγκόσμια. Τώρα, εμείς πάσαμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο πάτο. Το πιάσαμε πάτο. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς βλέπουμε ότι οι τιμές αυξάνονται αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να πούμε ότι οι αγορές δεν είναι σταθερές. Είναι ευαίσθητε, είναι ευπαθείς. Και κατά την απόψή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει γρήγορα να, απελευθερώσει, να απελευθερώσει αυτά τα αποθέματα παρέμβαση στην αγορά, αλλιώς η ισορροπία θα παρασαλευθεί. Τώρα, μέσα στην πραγματικότητα ενός γαλακτοκομικού τομέα, ο οποίο προσανατολίζεται περισσότερο προς την αγορά, είναι κάτι το οποίο μα βρήκε και εμά σύμφωνους, φυσικά η αστάθεια θα είναι ένα, μια σταθερά πολύ πιο παρούσα από ό,τι στο παρελθόν. Και σε κάποιο βαθμό η αστάθεια είναι κάτι το φυσιολογικό σε μια αγορά. Από την άλλη όμως, η υπερβολική αστάθεια και ρευστότητα συμφωνούμε όλοι μας ότι δεν είναι επιθυμητή είτε υπερβολικά χαμηλές τιμές είτε υπερβολικά ψηλές. Ακόμα και υπερβολικά ψηλές τιμές δεν είναι επιθυμητές, γιατί υπερβολικά ψηλές τιμές θα μπορούσαν να, να οδηγήσουν σε υψηλές τιμές για το ομό γάλα, για το ακατέργαστο γάλα. Το 2008 είδαμε ότι με αυτές τις ψηλές τιμές χάσαμε ε, και κέρδισαν οι ανταγωνιστές μας που δεν ασχολούνται με την παραγωγή γάλακτος. Δηλαδή, πολλοί πελάτες ε, πέρασαν σε πρωτεΐνες ε, που δεν προέρχονται από το γάλα. Επομένως και υπερβολικά υψηλές τιμές μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην αγορά. Τώρα, σε μια τέτοια ρευστή αγορά, μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου, ε, futures, ε, forward, ε, συμβόλαια κτλ. Αυτό μπορεί να γίνει μεταξύ των αγροτών και των συνεταιρισμών, ας πούμε, αλλά δεν θα μειώσει την ρευστότητα, θα περιορίσει τον κίνδυνο. Απλώς για τους εμπορευόμενους. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε, σε εθελοντική βάση. Αν ε, κοιτάξουμε την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το γαλακτοκομικό τομέα μετά το 2013, νομίζουμε ότι τα δημόσια εργαλεία μπορούν να μειώσουν, τα δημόσια μέσα μπορούν να μειώσουν αυτή την αστάθεια των τιμών. Και για να έχουμε ένα επίπεδο ασφαλείας όταν οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, ένα δίχτυ ασφαλείας, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση, ένα σύστημα παρέμβασης. Ίσως αυτό που έχουμε σήμερα για το γάλα και τη σκόνη γάλακτος και ιδιωτική αποθεματοποίηση. Όταν έχουμε χαμηλές τιμές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα futures Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν δίχτυ, ένα δίχτυ ασφαλείας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όμως και δημόσια μέσα με την διαχείριση των στρατηγικών αποθεμάτων. Ξέρουμε ότι σε φάση υψηλών τιμών μόνο τα τελευταία ε, κιλά ή τόνοι αποφασίζουν το πόσο ψηλές θα είναι οι τιμές. Μπορούμε να φανταστούμε ότι σε μια τέτοια κατάσταση η Κομισιόν στα πλαίσια της δυνατότητας διαχείρισης της αγοράς μπορεί να απελευθερώσει κάποιες ποσότητες από την αποθεματοποίηση. Επομένως θα πρέπει να έχουμε στρατηγική διαχείριση των αποθεμάτων. Αυτό πρέπει να κάνουμε όταν με ρωτάτε για το πώς θα διαχειριστούμε την αγορά στο μέλλον για να σταθεροποιήσουμε τις αγορές. Μια άλλη ερώτηση αφορά την ε, ιδιοκτησία των εταιριών που ανήκουν στην ΕΝΤΑ. Το 50% ε, ανήκει σε συνεταιρισμούς και το 50% των εταιριών είναι ιδιωτικές εταιρείες των εταιριών που ανήκουν σε εμά. Σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια, για τις σχέσεις τις συμβατικές μεταξύ των αγροτών και των, των συνεταιρισμών. Το 50% ε, της, της μεταποίησης γίνεται από συνεταιρισμούς. Νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά τα futures, ε, όλα αυτά τα μέσα, τα παράγωγα κτλ. να γίνονται εθελοντικά. Αυτή τη στιγμή ε, λειτουργούμε μέσα σε ένα πνεύμα που είναι πιο προσανατολισμένο προς την αγορά. Αν η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, περάσουν νομοθεσία για να επηρεάσουν τις συμβάσεις, τις τιμές, τους όγκους ε, μεταξύ των αγροτών και την ε, βιομηχανία, νομίζουμε ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει, δεν θα έπρεπε να επηρεάσει αυτή τη σχέση. Τώρα, για τον ΠΟΕ και την υποστήριξη του γαλακτοκομικού τομέα. Υπάρχει μια πρόταση επιτάπητος ε, στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ και οι τελευταίες προτάσεις κατά την απόψή μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις είναι το ανώτατο όριο στο οποίο θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε υπερβολικά πολλά. Τώρα ας κάνω και οι υπόλοιποι εταίροι και άλλοι τομείς κάτι ε, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι, θέλουμε να υπάρξει μια συμφωνία στον ΠΟΕ, γιατί πρέπει να εξάγουμε περίπου 8 με 9% της παραγωγής μας ε, προς τρίτες χώρες. Εάν δεν εξάγουμε αυτές τις ποσότητες σε τρίτες χώρες, τότε θα πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή μας κατά αντίστοιχα 8 με 9%. Ένας βουλευτής είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση στα σούπερ μάρκετ. και τι πρέπει να γίνει. Και τι πιστεύω εγώ για αυτήν την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειλικρινά, Πρόεδρε, έχουμε πολύ έντονο ανταγωνισμό στο εσωτερικό του γαλακτοκομικού τομέα. Και σε επίπεδο λιανεμπόρων επίσης υπάρχει ανταγωνισμός. Και σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ λιανεμπόρων και εκμεταλλεύσεων και συνεταιρισμών. Αυτή είναι η κατάσταση. Με το 2007 και το 2008 αυξήθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ των εμπόρων. Ε, είναι πολύ πιο έντονος από ό,τι πριν. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξετάσει την κατάσταση, να δει τι γίνεται με τις συμβάσεις, ε, με τα περιθώρια που έχουν, κέρδους που έχουν η βιομηχανία και για νέμποροι. Ε, γιατί όχι. Αλλά ο κλάδος χρειάζεται το λιανέμπορο και ο λιανέμπορος χρειάζεται τη βιομηχανία. Ένας βουλευτής είπε ότι οι τιμές του καταναλωτή παρέμειναν υψηλές και στο μεταξύ οι τιμές για τους παραγωγούς μειώθηκαν τότε το ερώτημα είναι ποιος, ποιος πήρε το κέρδος αυτό, ποιος το έβαλε στην τσέπη, ποιος καρπόθηκε αυτό το κέρδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλο το κέρδος πήγε στην τσέπη των λιανεμπόρων. Αν δεν ξέρετε ποια είναι η κατανομή αυτών των κερδών μεταξύ λιανεμπόρου και βιομηχανίας, δεν μπορείτε να απαντήσετε σωστά το ερώτημα αλλά θα μπορούσε κάλλιστα και η βιομηχανία να κέρδισε κάτι παραπάνω. Από αυτό το μεγαλύτερο κέντρο δηλαδή να πήρε κάτι παραπάνω. για τη διαφάνεια των τιμών. δεν είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στι τιμέ. Σε επίπεδο ε, εκμετάλλευση, ε, σε επίπεδο μεταποίηση, σε επίπεδο λιανεμπόρων. Για να σκεφτούμε λίγο τη διαφάνεια. Μήπως περισσότερη διαφάνεια θα ευνοούσε τους παραγωγούς ή θα ευνοούσε τους εμπόρους. Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί. Σίγουρα θα ξέχασα κάποια ερωτήματα, αγαπητέ Πρόεδρε, αλλά αυτά θέλω να απαντήσω σε μια πρώτη φάση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μπόκ. Ο κύριος Δράσμουσεν θα πάρει τον λόγο. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Thank you, Chairman. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, όπως συνήθως άλλωστε, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσα να διαιρέσω την εισήγησή μου σε δύο μέρη. Η πρώτη ενότητα είναι η γαλακτοκομική αγορά όσο έχει σήμερα. Και η δεύτερη η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εξέλιξη της. Η κατάσταση με τις τιμές ε, στην γαλακτοκομική αγορά, στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί δραματικά, τολμώ να πω, τους τελευταίους δύο μήνες. Δεν μπορούμε να κοφεύουμε στα πραγματικά στοιχεία οι τιμές για τη σκόνη, για τη τυριά, για το βούτυρο έχουν αυξηθεί. Και καιρός ήταν κιόλα. Έπρεπε να αυξηθούν. Και μάλιστα έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό. Προφανώς δεν στηρίζουμε πλέον με παρεμβάσεις στην κοινωτική αγορά. Αλλά σε τέτοιο βαθμό, επαναλαμβάνω, που την προηγούμενη εβδομάδα μειώσαμε όλες τις επιστροφές, εκτός από το βούτυρο. Για, όλες, για όλα τα άλλα προϊόντα μειώθηκαν σε μηδενικό επίπεδο. Και βλέπουμε ότι οι τιμές στην παγκόσμια αγορά, να σας δώσω ένα παράδειγμα, μια άλλη αύξηση ενός ηγετικού παραγωγιού της Νέας Ζηλανδίας της Νέας Ζηλανδίας αυξήθηκε για τη σκόνη γάλακτος κατά 15%. Άρα έχουμε μπει στην οδό προς την ε, σαφή και γρήγορη αύξηση των τιμών. Παρόμοια αύξηση τιμών όπως και το 2007. Σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί αυτή η τάση, κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να προβλέψει. στην παγκόσμια αγορά το θέμα είναι οι προπτικές παραγωγής στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία που αποτελούν σημαντικούς προμηθευτές παγκοσμίως εντός της κοινότητας. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει μία συνηθισμένη, αν θέλετε, καθυστέρηση μεταξύ των τιμών των πρώτων και των τιμών της μεταποιητικής βιομηχανίας, βλέπουμε αύξηση των τιμών της μεταποιητικής ε, βιομηχανίας στις βασικές χώρες παραγωγής. Και ναι, δεν αντιλέγω, ήταν χαμηλά τα επίπεδα. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Αλλά επίσης κανείς δεν αρνείται ότι το επίπεδο του 20 έως 30 λεπτών ανά το επίπεδο αυτό είναι πάνω από το επίπεδο που είχαμε πετύχει πριν από την ε, μεγάλη αστάθεια του 2007. Είναι επίπεδο υψηλότερο από τις ε, χρονιές του 2002-2006, όπου τα πράγματα ήταν ήρεμα. Τώρα το αναρκεί το επίπεδο αυτό των τιμών δεν μπορώ να το κρίνω εγώ τώρα, εδώ. Απλά διαπιστώνω ότι δεν μπορούμε να ασφαλίζουμε τα μάτια και να αρνούμαστε το γεγονός αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να στρεβλώσει αυτή την θετική εξέλιξη απελευθερώνοντας από θέματα το οποίο ανέφεραν πολλοί βουλευτές σήμερα βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι έχουμε σημαντική ευθύνη για την διαχείριση των αποθεμάτων. Και στο πλαίσιο αυτό να σας ε, πληροφορήσω κάτι. Να σας πω ότι μεγάλο τμήμα των αποθεμάτων αυτών παρέμβασης θα ε, χορηγηθεί μέσω του συστήματος ε, των πλέον απόρων, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ενώ στο παρελθόν μεγάλο τμήμα των ποσοστών παρέμβασης, των ε, αποθεμάτων παρέμβασης για το βούτυρο, για το γάλα το καθεξής μπορούσε να απελευθερωθεί άμεσα στο νέο σύστημα οι ποσότητες αυτές μπορούν να απελευθερωθούν μόνο από το Μάιο του 2010. Άρα δεν πρόκειται να απελευθερώσουμε τέτοια αποθέματα τους επόμενους έξι, μήνες. Και αυτό θα μας ε, επιτρέψει να δούμε μέχρι τότε αν η κατάσταση αυτή θα εξακολουθήσει να είναι σταθερή. Και ενδεχομένω, εάν αποδειχθεί ότι αυτό χρειάζεται, να απελευθερωθούν τα αποθέματα αυτά. Αλλά μόνο εφόσον χρειάζεται και μόνο με υπεύθυνο τρόπο όπως μας δώσει εντολή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά ως προς το τώρα, το σήμερα, αν θέλετε. Μέσα πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα άκουσα τις εισηγήσεις σας, ήταν πολύ επίκαιρες. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβω οποιαδήποτε δέσμευση πέρα από όσα ήδη κάνουμε. Έχουμε ιδρύσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου η οποία εξετάζει όλα αυτά τα θέματα τα οποία θίξονται σήμερα. Συναντήθηκε για πρώτη φορά η ομάδα εργασίας αυτή, είναι πολύ δραστηριά, συνεδριάζει πάλι αύριο και καλούμε τους βασικούς παράγοντες στην συνάντηση αυτή της ομάδας αύριο προκειμένου να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους εκπροσώπους των κρατών μελών τις δικές τους θέσεις, να παρουσιάσουν τη δική τους απόψη, να συμβουλεύσουν τις ομάδες αυτές. Διάφορες τέτοιες ενώσεις, όπως και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γαλακτοπαραγωγών. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή θα είναι πολύ χρήσιμη αύριο και η βάση της συζήτησης θα εστιαστεί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συμβατικές σχέσεις. Όλες, ε, όλων των ειδών τις συμβατικές σχέσεις. Πώς, πώς μπορεί να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών, γάλακτος, των εμπόρων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά και θα τα εξετάσει η ομάδα υψηλού επίπεδου. Επίσης το θέμα της διαφάνειας που ακούσαμε κάμποσες φορές σήμερα και αυτό θα τύχει εντελεχούς ανάλυσης στα πλαίσια της ομάδας υψηλού επίπεδου. Η ομάδα λοιπόν αυτή θα συναντηθεί, θα συναντηθεί τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μπορεί και δύο φορές. Αυτό θα καθοριστεί και από τις δυνατότητες που παρέχονται. Και σαφέστατα τα αποτελέσματα των ε, διαπραγματεύσεων θα συμπεριληφθούν σε σχετική έκθεση μέχρι τα τέλη του 2010. Πρόεδρε, ελπίζω να κατανοείτε ότι δεν ε, μπορώ να δεσμευτώ επί συγκεκριμένων στοιχείων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να το εξετάσουμε αυτό, όχι μόνο από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μία όσο πιο ευρεία εικόνα γίνεται αναφορικά με τον κλάδο της γαλακτοπαραγωγής μέχρι το τέλη του 2009 και ο σκοπός μας είναι να ταινίσουμε το μέλλον, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε από κοινού για να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση μέχρι το 2015 και πέρα από το 2015. Grazie. ευχαριστώ κύριε Ράσμουσεν. Και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Μπακ και όλους όσους έλαβαν μέρος σε αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση. Δεν λύσαμε φυσικά τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον εμβαθύναμε στην ανάλυση τους. Και στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα νέα προβλήματα που όπως διαπιστώσαμε θα γίνονται όλο και πιο συχνά στο μέλλον. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη έκθεση της ημερήσιας διάταξης που αφορά την πολιτική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και ποια είναι η ακολουθητέα στρατηγική. Έχουμε την έκθεση πρωτοβουλίας του κ. Τζανκάρλο Σκοτά. Είναι η δεύτερη φορά που εξετάζω αυτή την έκθεση. Η έκθεση του κ. Σκοτά δίνει μία απάντηση στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την πολιτική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων αφύπνισε το ενδιαφέρον χάρη και στις αρχικές διαβουλεύσεις ε, που έγιναν μετά την ε, υποβολή της Πράσινης Βίβλου. Πολλές ε, λύσεις δίνονται για τις γεωργραφικές ενδείξεις, για την πολιτική ποιότητα, για τις εμπορικές προδιαγραφές και τη βιολογική γεωργία. Ο εισηγητής θέλει να υπάρχει και μία νομοθεσία για την ετικητοθεσία πιο πλήρη ε, σύμφωνα με τα όσα προτείνει και η ίδια η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν επιπλέον όροι προαιρετικοί, ε, προϊόν ορεινό, ας πούμε, παράδειγματο χάρη προϊόν ε, με μικρή εκπομπή, χαμηλής εκπομπής άνθρακα. Ε, λοιπόν, τώρα θα πρέπει να δούμε ε, για τις τροπολογίες. Έχουμε προθεσμία μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 12 ε, η ώρα. Υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε την έκθεση την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, δηλαδή 1 και 2 Δεκεμβρίου. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σκοτά, ο οποίος θα μας παρουσιάσει εν συντομία το κείμενο της έκθεσής του. Υπενθυμίζω σε όλους τους συναδέλφους ότι στις 12 το μεσημέρι, 16 Νοεμβρίου, είναι τελευταία προθεσμία για τις απολογίες Και μετά την έκθεση ε, Σκοτά θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι παρόν ο κύριο Κορντονιέρ ε, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν συνεχεία θα πάρει το λόγο μετά τον κύριο Σκοτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι με την παγκοσμιοποίηση των αγορών και τη μεγάλη κρίση που ζει η Ευρώπη και στο γεωργικό τομέα, ε, μία από τις απαντήσεις που μπορεί να δώσει ο γεωργικός τομέας είναι να δώσει σημασία στην ποιότητα των προϊόντων. Θεωρώ ότι μια καλή ποιότητα μια καλή πολιτική ποιότητα ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και αυτό να αποτελέσει μια ε, προστιθέμενη αυξησει την ανταγωνιστικοτητα και αυτο να αποτελεσει μια προσθεμενη αξια για την οικονομία των ευρωπαϊκών περιφερειών, γιατί συχνά ε, για πολλέ ε, περιοχέ με περιορισμένε παραγωγικέ ικανότητε προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα ανάπτυξη. Η πολιτική συντομία της τη ποιότητα δεν μπορεί να διαχωριστεί από την υπόλοιπη κοινοτική γεωργική πολιτική, ούτε να αποσπαστεί από τι νέε προκλήσει όπω είναι η αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, η ανάγκη διατήρηση βιοπικιλότητα, ο ενεργειακό εφοδιασμό, η καλή διαχείριση των ζώων, ε, καθώ και η διαχείριση του νερού στη γεωργία, τομέα στον οποίο η κοινωνία απαιτεί βελτιώσει. Αυτά ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν τρία στοιχεία καταγραφής γεωγραφικών ενδείξεων. Ε, δείχνουν, υπάρχει μια σχέση με την πραγματικότητα που υπάρχει, εκπροσωπούν τις παραδόσεις, την ιστορία, το γούστο και τις αποκλειστικές γνώσεις που υπάρχουν για τα προϊόντα αυτά. Θεωρώ ότι και τα συστήματα ονομασίας προστατευόμενη προέλευσης και ειδική παραδοσιακά εγγυημένα προϊόντα, αυτά θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα. Ε, με αυτόν τον τρόπο ε, λαμβάνουμε υπόψη τη σχέση του προϊόντος και της ε, γεωγραφικής ε, ζώνης. Οι καταναλωτές συχνά μπερδεύουν την ε, ονομασία τόπου με την, ε, και δεν γνωρίζουν τη γνώση της διατροφικής αλυσίδας. Γι' αυτό θεωρώ ότι μόνο η υποχρεωτική ε, αναφορά του τόπου παραγωγής των πρωτογενών προϊόντων μπορεί να δώσουν στον καταναλωτή την πραγματική γνώση για την ποιότητα του προϊόντος που αγοράζει. Επίσης, ε, αυτό σε ένα, ε, υπόκειται σε ένα κύκλο παραγωγής, ο οποίος επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του, την ποιότητά του και την ασφάλεια τελικά και φυσικά τη διατροφική ασφάλεια. Άλλα δύο θέματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά και μπήκαν στην εκθεσή μου είναι η σημασία μιας ε, έντονης δράσης ε, εκπαίδευσης και ενημέρωσης ε, των καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν για τις εγγύησει των σημάτων, για τις εγγύησει και θα πρέπει να μπουν στα, στα διεθνή μητρώα και να αναγνωριστεί να αναγνωριστούν όλα αυτές οι γεωγραφικές ενδείξεις από το Παγκόσμιο Σύστημα του ΠΟΕ. Είναι η πρώτη μου έκθεση και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω επ' ευκαιρία τους ε, συναδέλφους. Θα κάνω λίγο λάθος την, παράγωγή την προφορά. Το Λέον Τζόρτζ, τον κύριο Ταμπάκη, ε, μάλλον ε, δεν τα είπα καλά τα ονόματά τους, και τον κύριο Λαβία. Ε, με τους οποίους συζητήσαμε αυτά τα θέματα. Τους ευχαριστώ για την ε, βοήθεια που μου έδωσαν, ε, για την σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριο Σκοτά. Και τώρα αρχίζει η συζήτηση. Ζήτησε το λόγο ο κύριος, η κυρία Γκαρσία. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Σκοτά για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Στο σχέδιο έκθεσης που μας υπέβαλε, περιλαμβάνει πολύ λογικά σημεία, πολύ εύστοχα και μπορούμε να τα ενσθενιστούμε. Για παράδειγμα, την δημιουργία ενός λογοτύπου ποιοτικών προϊόντων. Πιστεύω ότι αυτό το λογότυπο θα πρέπει να είναι απλό, φθηνό και για τα, να καλύπτει τα κοινοτικά προϊόντα. Γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιστοποιήσει την ποιότητα προϊόντων τρίτων χωρών. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι τρίτες χώρες στηρούν τις κοινοτικές προδιαγραφές και να τις ε, κατοχυρώνουμε το λογότυπο. Ο κύριος Κοτά μιλάει για την διατήρηση των, κανόνων ε, ε, των κοινοτικών κανόνων εμπορευματοποίησης. Μία υπερβολική απλούστευση θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε περισσότερα προβλήματα, όπως συμβαίνει με τα απορροκυπευτικά, που εξαιτία της υπεραπλούστευσης οδηγήθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν και άλλα σημεία όμως που θα πρέπει να επισημάνουμε από την έκθεση. Σε ό,τι αφορά την ενοποίηση των κανόνων για τις ε, ονομασίες προέλευσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, μείνει για το κρασί και για τα εινοπνευματόδη προστατευόμενη ονομασία προέλευση, γιατί η λειτουργία αυτών των κλάδων είναι πολύ διαφορετική και θα πρέπει να τύχουν ξεχωριστή ε, μεταχείριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μιλάει για την ενοποίηση των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών ενδείξεων, δεν μας δίνει σαφείς προτάσεις για το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η ενοποίηση. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε την εικόνα ποιότητας και την εντύπωση ποιότητας που δημιουργούν πολλά τέτοια κοινοτικά προϊόντα. Ο κύριος Κοτάκη που μιλάει για την προέλευση των πρώτων υλών, δεν θα πρέπει να αμελούμε και τις συνθήκες της βιομηχανίας. Το να επιβάλλουμε στη βιομηχανία την ένδειξη προέλευση των πρώτων υλών θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από λύσεις που θα φέρει για τον καταναλωτή. Δεν θα πρέπει να προσθέσουμε υποχρεώσεις ε, στην κοινωτική βιομηχανία, γιατί ήδη με την χρηματοπιστωτική κρίση και την υπερβολική γραφειοκρατία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ας μην τα επιτείνουμε εμείς με επιπλέον απαιτήσει. Επίσης, να γίνει μια περιπτωσιολογική ε, ανάλυση των κλάδων για να δούμε πού ε, μπορούμε να επιβάλλουμε τέτοια υποχρέωση και πού όχι. Ήταν πολύ στενή η συνεργασία που είχαμε με τον εισηγητή. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω ούτε να επαναλάβω κάποια θέματα που έδειξε ο κύριος Σκοτά. Θα ήθελα να πω ότι επί τη ευκαιρία της έκθεσης θα πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα το θέμα της ε, ολοκληρωμένης παραγωγής για να αξιοποιήσουμε την ποιότητα της κοινωτικής παραγωγής χάρη σε μια τέτοια ολοκληρωμένη παραγωγή. Θα φροντίσουμε να βοηθήσουμε τον εισηγητή για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως και ο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον κύριο Σκοτά με τον οποίο είχαμε πολύ ε, επικοδομητική συνεργασία και μάλιστα η ομάδα μας θα υποστηρίξει την έκθεση πρωτοβουλίας του. γιατί εστερνιζόμαστε τους τρεις στόχους της έκθεσης, δηλαδή την ε, δημιουργία ενός ε, περιεκτικού συστήματος ε, ε, μέτρων ε, ποιότητας της κοινοτική γεωργίας. Δεύτερον, χρειαζόμαστε πιο αξιόπιστες πληροφορίες και ταυτόχρονα θέλουμε μία απλοποίηση του συστήματος. Μερικές φορές υπάρχει αντίφαση μεταξύ του στόχου της απλοποίησης και της ανάγκης παροχής πιο αξιόπιστων πληροφοριών. Το πρώτο θέμα αφορά το κοινοτικό λογότυπο. Εμείς είμαστε υπέρα του κοινοτικού λογοτύπου, του λογοτύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνούμε με την πρόταση του εισηγητού να μην έχουμε δεύτερο και δεύτερο κοινοτικό λογότυπο. Γιατί όπως θα θυμάστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει και την εισαγωγή και δεύτερου λογότυπου ΕΕ για μη ε, κοινοτικά προϊόντα που πληρούν όμως τις κοινοτικές προδιαγραφές ε, γεωργικής παραγωγής. Αλλά συμφωνώ με τον εισηγητή και είμαι και εγώ κατά της εισαγωγής δεύτερου λογοτύπου. Σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμφωνώ με τον εισηγητή, γιατί για τις παλιές χώρες μέλη η διαφοροποίηση μεταξύ προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ε, και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ε, δεν υπάρχει. Σεβόμαστε βέβαια τις πρακτικές και τις απαιτήσει των παλιών χωρών μελών που έχουν αυτή τη διαφοροποίηση που στις νέες χώρες δεν υπάρχει και επίσης ε, συμφωνούμε με τη διατήρηση του ισχύοντος συστήματος και συμφωνούμε με τον ε, εισηγητή. Για τον Ίνο, ο... στη Γαλλία η κουλτούρα της κατανάλωσης κρασιού είναι πολύ υψηλή και ο καταναλωτής είναι πολύ απαιτητικός. Βέβαια, πολλέ φορέ δεν γίνεται διάκριση μεταξύ του ΠΟΠ και του πήγαμα ε. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι το σύστημα θα πρέπει να μείνει αμετάβλητο. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό λογότυπο για τη βιολογική γεωργία, θα πρέπει να γίνει μια ενοποίηση εδώ, γιατί με την παρούσα κατάσταση παρακολύεται ουσιαστικά η κοινοτική βιολογική γεωργία και το διακρατικό εμπόριο βιολογικών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά το εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι το σύστημα θα πρέπει να διασφαλιστεί και δεν συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει κατάργηση του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, παρόλο που το σύστημα είναι σχετικά καινούριο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σύστημα, αλλά να αποσαφινιστούν οι συνθήκες καταχώρησης για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά το, τη χαμηλή εκπομπή άνθρακα ή το αποτύπωμα άνθρακα, πιστεύω ότι αυτό το αποτύπωμα άνθρακα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα τρόφιμα. Είμαι υπέρ του υποχρεωτικού, του δεσμευτικού χαρακτήρα του αποτυπώματος διοξιδίου του άνθρακα για τα τρόφιμα. Επίσης, Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειαζόμαστε μία συνολική ενημερωτική εκστρατεία ή εκστρατεία διαπαιδαγώγησης του κοινού. Θα πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα τον καταναλωτή για πολλά θέματα και για τους καταναλωτές οι γραμμικοί κώδικες και οι πληροφορίες από την ιστοσελίδα μπορούν να, να πλουτίσουν την ενημέρωσή του χωρίς ταυτόχρονα να επιβάλλουν ε, την ε, ε, αύξηση των πληροφοριών στα ίδια τα τρόφιμα. Χάρη στους γραμμικούς κώδικες και στη ριστοσελίδα μπορούμε να έχουμε πλούσια και αξιόπιστη πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Σεγετά. Ευχαριστώ τον κύριο Ταμπάτσι. Καρσία Πέρες. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σκοτά για την έκθεσή του και σίγουρα συμφωνούμε όλοι για την ανάγκη ποιότητας της κοινοτικής παραγωγής. Θα ήθελα να επενέσω τον εισηγητή για την έμφαση που δίνει στην ανάγκη προαγωγής των κοινοτικών προϊόντων και στην ενημέρωση. Χρειαζόμαστε καλύτερη παγκόσμια προστασία για τις γεωγραφικές ενδείξεις και ένα κοινοτικό λογότυπο για τη βιολογική γεωργία. Η ενίσχυση της ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής και των χαρακτηριστικών ποιότητας των γεωργικών προϊόντων είναι πολύ σημαντικό και ωφελεί την ύπεθρο γιατί όχι μόνο θα βελτιώσει το γεωργικό εισόδημα αλλά ταυτόχρονα θα σταθεροποιήσει τον πληθυσμό στην ύπεθρο γιατί πολύ συχνά υπάρχει ε, αστιφιλία και έξοδος από τις γεωργικές περιοχές εξαιτίας των δεινών ε, συνθήκων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προωθήσουμε αυτή την πολιτική ποιότητα. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες εμπορευματοποίησης, σίγουρα η απλούστευση θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της ενημέρωσης του καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά την σήμανση της προέλευσης θα πρέπει να συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία για τη σήμανση και να εξεταστεί περιπτωσιολογικά για να αποφευθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τι τις διάφορες ενδείξεις διαφοροποιημένης ποιότητας που υπάρχει σε κοινοτικό επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια έχουμε διάσταση απόψεων με τον εισηγητή, αλλά πιστεύω ότι στη διάρκεια της εξέτασης αυτής της έκθεσης θα καταλήξουμε σε, συμβα... σε σημαντικές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Σίγητα, θεωρώ ότι το έγγραφο είναι πάρα πολύ καλό. Ωστόσο θα ήθελα να γίνουν λίγο πιο έντονα διακριτά κάποια στοιχεία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Το γεγονός δηλαδή ότι θα πρέπει να τριθούν οι παραδόσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό για όσους θέλουν να διατηρηθεί ζωντανή η πολιτισμική, πολιτισμική κληρονομιά της υπαίθρου. Θα πρέπει να προστατεύσουμε και την πολιτιστική κληρονομιά αυτή. Και υπάρχει άλλο ένα στοιχείο. Το γεγονός ότι η σύγχρονη βιομηχανία και η βιομηχανία τροφίμων έχει ψηφιοποιηθεί πλέον. Ποιος λοιπόν θα συνεχίσει στο μέλλον την ε, παραγωγή τροφίμων, όταν όλα πλέον θα γίνονται με υπολογιστές. Ποιος θα ψήνει το ψωμί. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την ε, παραδοσιακή κληρονομιά. Γι' αυτό λοιπόν στο σημείο αυτό επιθυμώ να διατυπωθεί πιο έντονα το κείμενο στη συνέχεια. Δύο παρατηρήσεις οι οποίες μπορεί να σας ακούγονται κάποιες παράλογες. Ελπίζω λοιπόν σωστά να σας τα εξηγήσω. Όταν μιλάμε για την επισήμανση των τροφίμων και για την μεγαλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή, αυτό που θα καταλήξει σε μία ατελείωτη γκάμα επισημάνσεων για όλα τα τρόφιμα, για τον τρόπο παραγωγής, την προέλευση, την παραδοσιακή αξία τους. Πόσες επισημάνσεις πια θα συζητηθούν στην... Ε, πόσα σήματα θα συζητηθούν πια. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παραγωγή θα πρέπει να γράφουν πάντα, να αναγράφουν τις ε, σημάνσεις, τα σήματα που επιθυμούν, αλλά θα πρέπει να μην προκαλούν σύγχυση του καταναλωτή, να μην παραπλανούν τον καταναλωτή. Μπορεί κανείς να γράψει ό,τι θέλει, αρκεί να το αποδεικνύει. Αν για παράδειγμα, εγώ παράγω λουκάνικα, ας πούμε, και λέω ότι το κρέας αυτό προέρχεται από εξαιρετικά ευτυχισμένα ε, γουρούνια. Πρέπει να το αποδεικνύω αυτό. Να αποδείξω ότι η χείρη μου όντω είναι πιο ευτυχισμένη από άλλου χείρου. Ναι, με συγχωρείτε για το παράδειγμα, αλλά προ αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να κινηθούμε. Να τηρηθούν κάποιες αρχές και να τι ορίσουμε τις αρχές αυτές για να μην καταλήξουμε να έχουμε τριών χιλιάδων διαφορετικά σήματα. Κάτι άλλο τώρα κατά την εμπορία, για παράδειγμα, των ε, ηχθείων ηχθειοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι δεν καλλιεργούνται τα ψάρια. Πρόκειται για ένα προϊόν ζωντανό, από ζωντανούς οικοτόπους, από τις ακτές. Όταν πολλούνται τα ψάρια αυτά, εχθειοκαλλιέργειες. Αγοράζοντας ε, ψάρια εχθειοκαλλιέργειας, ε, ουσιαστικά τι κάνουμε, ε, γλιτώνουμε τα ψάρια της θάλασσας. Αυτό είναι τελείως παράλογο, γιατί τα ψάρια αυτά στοιχίζουν 3, 3 έως 5 ε, ψάρια τη ανοιχτή θάλασσα. Δηλαδή, αυτό κάπου δεν πρέπει να αναφέρεται ότι όσο πιο πολλά ψάρια χθιοκαλλιεργείς καταναλώνουμε, τόσο πιο πολλά ψάρια χάνουμε από την ελεύθερη θάλασσα. Ευχαριστώ κυρία Πόλσον. Ε, τώρα η κυρία Ντελάνζο. Κύριε Τελάμε, να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και σας εισηγητά για την εισαγωγή σας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η έκθεση. Το πιο σημαντικό που θέλουμε ως Επιτροπή είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας και αυτό θα είναι αρκετά δύσκολο γιατί βλέπω ότι γίνεται και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε και νομίζω ότι θα έχουμε πολλή δουλειά για να πείσουμε όλο το Κοινοβούλιο. Κάποια άλλα στοιχεία τώρα σε ό,τι αφορά τις επιπλέον, ε, τα επιπλέον σήματα στην ετικέτα να σας πω με πάσα ειλικρίνεια ότι αντιμετωπίζω την εξής πρόκληση. Καταρχάς τους ορισμούς. Φυσικά είναι καλύτερο να υπάρχουν ευρωπαϊκοί ορισμοί, για παράδειγμα, για το αποτύπωμα της, ε, του άνθρακα. Αυτά που προβάλλει, για παράδειγμα, μία σειρά σούπερ μάρκετ στην Αγγλία δεν με πείθουν, δεν σημαίνουν τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ευρωπαϊκοί ορισμοί σε συνεργασία με τον κλάδο για να δούμε τι θα σημαίνουν αυτοί οι ορισμοί. Αλλά αφετέρου υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία παίζουν μεγαλύτερο ρόλο σε κάποια κρατημέλη από ότι σε άλλα. Για παράδειγμα, όταν, για παράδειγμα, ζω σε ένα κράτος μέλος όπου ζει έξι μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, ε, δεν μας ενδιαφέρει πολύ τι γίνεται με την ορεινή καλλιέργεια, αλλά αυτό που απασχολεί την Ολλανδία, για παράδειγμα, είναι η παραγωγή γάλακτος. Αν προέρχεται από αγελάδες οι οποίες βοσκούν ελεύθερες όλο το χρόνο και όχι από αγελάδες εκτροφής. Αυτό μπορεί να απασχολεί λιγοτερα άλλα κρατημέλη. Πόσο λοιπόν θα πρέπει να περιορίσουμε και θα πρέπει να καθορίσουμε ε, στα κράτη-μέλη ποια σήματα θα χρησιμοποιήσουν, μήπως καλύτερα να αποφασίσουν τα ίδια μόνα τους, ε, τι χρειάζεται για το κάθε κράτος μέλος. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα συνεννοηθούμε σωστά. Κάποιες άλλες μικρές παρατηρήσεις. Δεν συμφωνώ με μια έκθεση που αναφέρεται, με μια έκφραση που αναφέρεται στην έκθεση, ότι πρέπει να περιλαμβάνονται όσο πιο πολλές πληροφορίες γίνεται στην ετικέτα. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν είναι η ετικέτα ο τρόπος πληροφόρησης του καταναλωτή. Είναι περιορισμένος ο χώρος που έχει η ετικέτα τέτοια θέματα, για παράδειγμα στοιχεία όπως ε, η προέλευση, η τοποθεσία του αγροκτήματος. Μήπως θα πρέπει να μπουν όλα αυτά στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, σήμερα μπορούμε να δούμε από πού προέρχεται ε, το ζώο, πότε γεννήθηκε, πότε καταναλώθηκε. Όλα αυτά νομίζω χρειάζονται και χρειάζονται πιο πολλές πληροφορίες πέρα από τις πληροφορίες που χωράνε σε μια ετικέτα για τον βιολογικό λογότυπο θα υποβάλω και τροπολογία ε, για τον πιο αυστηρό έλεγχο των βιολογικών προϊόντων γιατί όλα ξεκινούν και τελειώνουν στον έλεγχο τη στιγμή που τα προϊόντα φεύγουν ή μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές το έχουμε συζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζονται πιο πολλά χρήματα για τους ελέγχους και σίγουρα θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίες. Αλλά σε γενικέ γραμμές πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόταση του εισηγητή. E Κύριος Λαβία τώρα και μετά ο Όρφων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Σκοτά για αυτή την εισαγωγική παρουσίαση που μας έκανε, την οποία συμφωνώ πλήρως, ε, ιδίως ό,τι αφορά την διάκριση των συστημάτων ποιοτικής ε, εξασφάλισης και το περιεχόμενό τους. Τώρα, βεβαίως μπορούμε να εμβαθύνουμε στους όρους και να φτάσουμε σε καλύτερο ορισμό ε, μέσα από συζήτηση στο εσωτερικό της Επιτροπής μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε για τους επιπρόσθετους όρους. Ε, αυτό που είπε μάλιστα και ένας συνάδελφος για, τις, ε, για διάφορες παραγωγές, που είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης, που δεν χρησιμοποιείται ακόμα πολύ στην, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ακόμη περισσότερο κάποια στοιχεία που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Το θέμα της επικοινωνίας που είπαν πάρα πολύ. Ε, έχει μεγάλη σημασία. Σε ορισμένε ε, περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι τα δύο τρία των καταναλωτών δεν γνωρίζουν τη σημασία των επισημάσεων σε ό,τι αφορά αυτά τα συστήματα ποιότητας. Επομένως, δεν έχει νόημα να βασίσουμε την ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική ανταγωνιστικότητα, αν οι καταναλωτέ δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το περιεχόμενο και το σύμβολο που υπάρχει σε ετικέτε. Νομίζω ότι οι πολιτικές επικοινωνία θα πρέπει να ενδυναμωθούν ε, και να, τονιστού, να τονιστεί ότι στα προγράμματα του δεύτερου πυλώνα, όπως σήμερα προβλέ... κάτι που προβλέπεται μόνο μερικά σήμερα, θα πρέπει και για τους ιδιώτες και για τους συνεταιρισμούς ε, να μπορούν μαζί να κάνουν ε, εκστατείες επικοινωνίας ε, με κονδύλια και των διαρθωτικών ταμείων για τα σήματα, ούτως ώστε να δίνουν περισσότερες πληροφορίες και να αφυπνιστούν οι καταναλωτές. Ευχαριστώ τον κύριο Δηλαδή, τώρα ο κύριος Ντόρφμαν. Και συνεχεία κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση του συναδέλφου Σκοτά είναι πάρα πολύ καλή και είναι και πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της γεωργίας. Δύο στοιχεία ήθελα να θίξω. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν το θέμα της ε, προέλευσης της πρώτης ύλη. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι μόνο να δώσουμε τις σωστές πληροφορίες στον καταναλωτή, αλλά να δούμε και πού είναι η προστιθέμενη αξία της παραγωγής αυτής γιατί είμαστε Επιτροπή Γεωργίας και είμαστε υπεύθυνοι να διασφαλίσουμε η υπεραξία αυτή να μην περιοριστεί στη βιομηχανία αλλά και στον αγρότη. Και νομίζω ότι πολλά προϊόντα σήμερα, για παράδειγμα στον κλάδο του κρέατος, όπου η προέλευση του κρέατος δεν αναφέρεται και η προστιθέμενη αξία ε, έγινε μόνο στην βιομηχανία. Ο αγρότης δεν κερδίζει τίποτα γιατί η πρώτη ύλη δεν αναγνωρίζεται. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε προκειμένου να υποφελούνται και οι γεωργοί και οι εκμεταλλευτές. Δεύτερο στοιχείο που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, το θέμα της φορολόγησης προσφοράς. Μάλλον, συγγνώμη, της ε, ε, διαμόρφωσης της προσφοράς. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να ελέγξουμε και το θέμα της προσφοράς. Εδώ εισέρχεται ένα στοιχείο διαεπαγγελματικών ε, σχέσεων. Και υπάρχουν πολλά εξαιρετικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να διαμορφωθούν ε, και να διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο οι τιμές ενός προϊόντος. Αυτό εξαρτάται από την ποσότητα που διατίθεται στην αγορά. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε λοιπόν αυτό το στοιχείο. Και τέλος ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σκοτά για τη ρητή αναφορά των ορεινών περιοχών στην έκθεσή του. Αιούζο, εντόπο... Αιούζο και μετά Ντάντα. Ευχαριστώ. gracias, señor θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους και εισηγητές για το έργο τους και τις παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Εγώ θα συντάξω τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό και θα ήθελα να πω ότι στην Ευρώπη έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες για την ποιότητα και την παραγωγή τροφίμων. Οι κανόνες αυτοί είναι πολύ ανώτεροι από αυτούς που ισχύουν στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τα κοινοτικά προϊόντα να χαίρουν ξεχωριστού λογοτύπου για να γνωρίζουν οι καταναλωτέ ότι αυτό που αγοράζουν είναι τρόφιμο που παρήχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώντας τις αυστηρές προδιαγραφές που ισχύουν εδώ. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο υπόλοιπο κόσμο δεν είναι τόσο απαιτητικό. Και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις προδιαγραφές των τρίτων χωρών, είναι αδύνατον. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κοινοτικό λογότυπο σε εξωκοινοτικά προϊόντα. Οι ονομασίες προέλευσης και οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις επίσης είναι ίδιων της κοινοτικής ποιότητας και δίνουν προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και τις δύο κατηγορίες. Μέχρι στιγμής απέδειξαν την εύρυθμη λειτουργία τους και στον Ίνο όπου ισχύει ε, μία από τις παλιότερες προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης. Δεν θα πρέπει να υποβαθμίσουμε τους κανόνες για να επιτρέψουμε νέες γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης, γιατί έτσι θα υποβαθμίσουμε τα συστήματα αυτά. Τέλος, η σήμανση και η ευρωπαϊκή σήμανση θα πρέπει να είναι ενιαία, μία και μόνο, και η σήμασή αυτή θα πρέπει να είναι ενιαία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ενιαία είναι και οι κανόνες που ισχύουν και οι προδιαγραφές. Και επιπλέον θα μπορούσε να αναφέρεται και η ένδειξη τόπου παραγωγής πρώτων υλών. Θα πρέπει τα πράγματα να είναι απλά και εύκολα, γιατί αν τα περιπλέξουμε το σύστημα θα γίνει ανέφικτο και ανεφάρμοστο. Και μετά Ζωζέ Μποβέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ποιότητα της δουλειάς του και την ικανότητα υπομονή, και την υπομονή του όταν του διατυπώναμε κάποιες προτάσεις. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Στις διάφορες ανακοινώσεις της Επιτρόπου ή των υπηρεσιών της Επιτροπής για αυτό το θέμα, η Κομισιόν προβλέπει να κατακαιρματίσει, να το πω έτσι, την διαδικασία πιστοποίησης ούτω ώστε να κρατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο απλώ κάποια προϊόντα τα οποία πηγαίνουν και σε ξένε αγορέ. Αυτό το θέμα νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν αναφέρεται στην έκθεση. Νομίζω όμω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρει θέση για αυτό το θέμα. Το να κατακαιρματίσουμε τη διαδικασία πιστοποίηση νομίζω ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγχυση αύριο μεθαύριο στο πνεύμα των καταναλωτών. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε μια ενιαία διαδικασία αναγνώρισης των διαφόρων λογοτύπων μας. Ευχαριστώ. Ζωσέ Μποβέ και εν συνεχεία κυρία Μαγκίνες. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε και να κάνω κάποιες διευκρινήσεις ε, ή να ζητήσω διευκρινήσεις για το σημείο 6, 7, 8, 16 και 26. Είναι πολύ συγκεκριμένα λοιπόν αυτά που θέλω να ρωτήσω και δεν θέλω να δημιουργήσω πολεμικέ. Το πρώτο θέμα, ε, και δεν θα επανέλθω, είναι το θέμα ε, ποιότητα Παύλα Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα, αντίθετα από αυτό που ακούστηκε από ένα συνάδελφο, ε, φοβάμαι ότι θα δημιουργηθεί σύγχυση ε, με τα πραγματικά σήματα ποιότητα γιατί δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή, ένας ευρωπαϊκός κανόνας παραγωγής. Εκτός και να αποφασίσουμε να καθορίσουμε ένα πλαίσιο για τους κανόνες παραγωγής, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στο βαθμό που δεν υπάρχει θα δημιουργήσουμε σύγχυση. Στο σημείο 7 της έκθεσης, για τους κανόνες εμπορευματοποίησης ε, και τα πρότυπα εμπορίας. Θα πρέπει να παραμείνουμε σε μια λογική έτσι, ενός προτύπου κλασικού ή να προβλέψουμε μια επέκταση σε, σε κάποιες άλλες ε, σε κάποιες άλλες δυνατότητες, όχι τόσο τυποποιημένες, που θα δείχνουν και την ποικιλομορφία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομίζω ότι εδώ κάτι θα πρέπει να προσθέσουμε, κάποια διευκρίνηση θα πρέπει να κάνουμε. Στο σημείο 8, για το θέμα των, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης. Το θέμα που τίθεται είναι ο καλύτερος οργανισμός για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δεν θα πρέπει καλύτερα να επανέλθουμε ε, στις, σε αυτό που υπάρχει εδώ σε επίπεδο υπηρεσιών, στις αζώνες δηλαδή. Γιατί νομίζω ότι ο δημόσιος έλεγχος εκεί γίνεται καλύτερα. Για το θέμα της αξιολόγησης συμφωνώ πάρα πολύ ε, καλά. Νομίζω ότι πρέπει, πρέπει να έχουμε πραγματικά εργαλεία για να μην υπάρχουν απάτες ε, ούτω ώστε να μην ε, έχουμε προϊόντα τα οποία μιμούνται τι ονομασίε προστατευόμενη προέλευση και τη προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Στο σημείο 26 τώρα λέμε ότι θα πρέπει να καταγράφουμε τη χώρα προέλευση. Θα πρέπει να πάμε πιο μακριά. Θα πρέπει να υπάρχει μια ένδειξη, ούτω ώστε να υπάρχει διαφάνεια για τον καταναλωτή σε ό,τι αφορά την προέλευση του προϊόντος. Ευχαριστώ, Ζωζέ. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Να ρωτήσω τον εισηγητή, εάν κοίταξε τις επισημάνσεις όπου συχνά ε, ο κόσμος, ε, ξέρετε, ότι βγαίνει συχνά έξω από το σπίτι του, δεν, δεν τρώει μόνο στο σπίτι, τρώει σε εστιατόρια κτλ. Ε, μπορούμε να ξέρουμε από πού ε, προέρχεται το κρασί αλλά συχνά οι πρωτεΐνες, το κρέας και τα λοιπά που τρώμε έξω από το σπίτι μας, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Οπότε τι γίνεται με αυτή την ενημέρωση. Ε, κλείνουμε τις παρεμβάσεις ε, με τον κύριο Σεκερέσκι. Και... μετά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαι λακωνικός. Έχω μία ερώτηση προς τον εισηγητή σας και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί, γιατί είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία της καταχώρησης μερικές φορές κρατάει μέχρι και τρία χρόνια. Είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο. Δεύτερο πρόβλημα. Τι δυνατότητες υπάρχουν και τι όροι στήριξη στο μέλλον για τα παραδοσιακά προϊόντα, για τα παραδοσιακά τρόφιμα ή για τα προϊόντα τα βιοτεχνικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη αυτών των εγκυμένων παραδοσιακών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά την προέλευση της πρώτης ύλη και του κόστους, στην περίπτωση του γάλακτος, ας πούμε, έχουμε την τιμή των ε, ζωοτροφών που επηρεάζουν την τιμή του γάλακτος. Το ίδιο και στα άλλα τρόφιμα υπάρχουν και συναφή κόστη που επηρεάζουν την διαμόρφωση μιας τιμής. Γιατί σίγουρα η προέλευση των πρώτων υλών και η τιμή των πρώτων υλών επηρεάζουν και την τιμή του τελικού προϊόντος, αλλά και τη γεύση πολλές φορές. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Κορμπενιέ, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συνεχεία στον εισηγητή που θα απαντήσει στι ερωτήσει που έγιναν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, εξαιρετική του έκθεση και την προσπάθεια που έκανε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται ιδιαίτερος ε, για την υποστήριξη που έδειξε ο συγητής προς την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλά στοιχεία της ανακοίνωσης υποστηρίζονται σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Επίσης, ε, συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους, ως προς την ανακοίνωση αλλά και ως προς το τι μελιγενέστε. Γιατί θα ακολουθήσουν ε, νομοθετικές προτάσεις κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διεκπαιρεωθεί αυτή η διαδικασία. Έχω ορισμένε παρατηρήσεις και ελπίζω να ικανοποιήσω την περιέργεια πολλών ε, που έθεσαν ερωτήσεις. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό λογότυπο, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ένα στοιχείο για το λογότυπο αυτό. Αυτό το λογότυπο ευρωπαϊκής ποιότητας είναι ένα θέμα που συζητάται χρόνια ολόκληρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, διαλεκτική και πολύ ανοιχτή ως προς την ιδέα αυτή. Τελικά απέκλεισε αυτή τη δυνατότητα, όπως φαίνεται και στην ανακοίνωση, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από τους πρωταρχικούς λόγους πάντως ήταν ότι όλες οι διαφερόμενες πλευρές αντιτάχθηκαν σε αυτή την ιδέα στη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την πράσινη βίβλο. Κανένας δεν υποστήριξε αυτό το λογότυπο, γιατί το λογότυπο ε, εγγυάται μόνο τους ε, κανόνες ε, γεωργικής κοινοτικής παραγωγής και δεν είναι... Ε, και σε τέτοια περίπτωση ήταν ανοιχτό και για όλα τα εξωκρατικά προϊόντα που τηρούσαν τους ίδιους ε, κανόνες και προδιαγραφές. Κάτι τέτοιο όμως θα δημιούργησε σύγχυση για τον καταναλωτή. Γι' αυτό όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές ε, τάχθηκαν κατά του λογοτύπου. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίμησε να προτείνει την ένδειξη του, του τόπου παραγωγής. Κάτι που βρίσκει σύμφωνο και τον εισηγητή. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα ποιότητας, προστατευόμενη ονομασία προέλευση και γεωγραφικών ενδείξεων, Καταρχήν για τα τρία μητρώα. Πρότασή μας ήταν να απλουστευτεί το σύστημα γιατί υπήρχαν διαφορετικά μητρώα και διαφορετικές βάσεις δεδομένων, αλλά και διαφορετικές περίοδοι για την υποβολή ενστάσεων. Υπάρχει δυνατότητα απλοποίησης του συστήματος για να είναι πιο εύχριστο και πιο σαφές και πιο εύληπτο σε μια κοινοτική νομοθεσία που θα συγκεντρώσει τα κοινά στοιχεία και θα προβεί σε μια εναρμόνιση όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Βέβαια δεν θέλουμε να ισοπεδώσουμε τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων παραγωγών και προϊόντων, για παράδειγμα του ίνου, των ινοπνευματοδών ή των άλλων γεωργικών προϊόντων. Τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε παραγωγής θα προστατευτούν. Και θέλουμε να υπολογίζουμε και στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση αυτή. Σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση των προστατευόμενων ονομασιών προέλευση και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, η ανακοίνωσή μας ε, αναφέρει ως πιθανή αυτή την ε, πρώτη λύση. Θα εξεταστεί λοιπόν αυτή η δυνατότητα συγχώνευσης ε, των ΠΟΠ και πήγαμε ε, αλλά επί του παρόντος δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά. Σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα, τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, διαπιστώνω ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την πρόταση αυτή. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προωθήσει αυτά τα προϊόντα, να αναδείξει την αξία τους και να τα προαγάγει. Γι' αυτό και μιλήσαμε για την πρόταση των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων. Γιατί σήμερα έχουμε καταχωρημένα περίπου 20 προϊόντα στην κατηγορία αυτή την τελευταία 20 ετία. Γι' αυτό και θεωρούμε το σύστημα όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Σίγουρα θα υπάρξει ένας καλύτερος τρόπος για την πρόωθηση των παραδοσιακών σπεσιαλιτέ. Και αυτόν τον τρόπο θα αναζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο τελευταίο σημείο της ανακοίνωσης που μιλά για τα ιδιωτικά συστήματα πιστοποίησης. Τα συστήματα αυτά ε, γνώρισαν εκθετική αύξηση τα τελευταία χρόνια αλλά ίσως δημιουργούσαν προβλήματα και επιπλέον κόστος για τους παραγωγούς. Άλλωστε ενέχουν και τον κίνδυνο σύγχυση για τους καταναλωτές. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι θα πρέπει να περιορίσει τα προβλήματα από τα συστήματα αυτά, αν και δεν κρίνει σκόπιμο προς το παρόν να καταθέσει νομοθετική πρόταση για το θέμα αυτό. Προτιμά να υποβάλει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας αναπτύξει από κοινού με τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Τέλος, για τις διαδικασίες καταχώρησης, που ήταν μία από τις ερωτήσεις, έχουμε επίγνωση της βραδύτητας ε, και της ε, μεγάλης διάρκειας αυτών των διαδικασιών, γιατί γίνεται μια πρώτη ανάλυση σε εθνικό επίπεδο και κατόπιν δεύτερη ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει η δέσμευση να δοθεί μια απάντηση ήδη από το πρώτο έτος, δηλαδή το πολύ 12 μήνες μετά την λήψη της αίτηση από το κράτος μέλος. Αυτή είναι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει μέσα σε ένα χρόνο. Και στην ανακοίνωση αναλαμβάνουμε και τη δέσμευση να επιταχύνουμε περαιτέρω τις διαδικασίες μελέτης αυτών των ετοιμάτων και την λήψη απόφασης ως προς τις αιτήσει που υποβάλλονται. Και μάλιστα μερικές φορές θα απορρίψουμε και κάποιες αιτήσει που δεν τις κρίνουμε ικανοποιητικέ. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Κορδονιέ. Και τώρα ο Τζαν Κάρλο Σκοτά θα δώσει κάποιες ε, απαντήσεις και θα διευκρινίσει κάποια πράγματα. επαναλαμβάνω στους αδέλφους ότι θα πρέπει να υποβάλουν τις τροπολογίες τους μέχρι τις 16 του μηνός, 12 η ώρα το μεσημέρι και θα εγκρίνουμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής την ε, έκθεση αυτή 1η ε, Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Από αυτά που άκουσα, είναι μια έκθεση η οποία προκύπτει από σύγκληση των απόψεων των ανθρώπων που συναντηθήκαμε και συζητήσαμε. Δηλαδή, ακούστηκαν πολλέ ιδέες ε, και πολλά χέρια έγραψαν αυτή την έκθεση. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το λογότυπο ποιότητας, ε, το οποίο καθορίζει και εξασφαλίζει την ασφάλεια του προϊόντος και καθησυχάζει το πνεύμα του καταναλωτή. Γι' αυτό σκεφτήκαμε αυτό το λογότυπο. για να προωθήσουμε αυτή τη δουλειά που κάνουν οι παραγωγοί μας και το ότι κάνουν ποιοτικό προϊόν ε, μέσα από ένα λογότυπο που εξασφαλίζει στους καταναλωτές ότι το προϊόν παράγεται στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Καλή ιδέα αυτή για την ποικιλομορφία ε, της παραγωγής, ε, ότι η παραγωγή δεν γίνεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά υπάρχουν πολλές συνιστώσεις, θα πρέπει να το αναφέρω. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. Ακούστηκαν και άλλες ιδέες, αλλά αυτή είναι η ιδέα που συνάντησε τη μεγαλύτερη συνένεση. Ακόμη και εθνικές ε, δημόσιες αρχές ελέγχου θα μπορούσε να είναι μια ιδέα για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στα προϊόντα. Ευχαριστώντας όλους, θα ήθελα να σας πω κάτι πραγματικά ειλικρινές. Σημειώνω αυτά τα χρόνια ότι η αλλαγή του τρόπου παραγωγής, η αλλαγή των πρακτικών της γεωργίας, η εγκατάλειψη κάποιων ζωνών, ακριβώς αυτές που προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε, άλλαξαν τη, τη, τη φύση του τοπίου μας και όχι προς το καλύτερο κατά, ανάγκη. Νομίζω ότι η ιστορία μας, η κουλτούρα μας, ο, η μέθοδος που χρησιμοποιούσαμε για την παραγωγή θα πρέπει να διατηρηθεί. Γιατί χάρη σε αυτή τη διατήρηση θα ελέγξουμε το, το, τη γη μας. Όπως οι, οι παλιοί ξέρανε με τέσσερις πέτρες και λίγη γη να φτιάξουν ε, ένα προϊόν η όψη της υπαίθρου, η επιστροφή του κόσμου και κυρίως των τουριστών ε, σε αυτά τα μέρη. Ε, αυτά τα, αυτοί οι μικροί θύλακες ε, ποιότητας ε, στα βουνά μας, σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές, είναι στοιχεία ποιότητας τα οποία με, για μένα είναι πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ για τις θέσεις σας. Αν έχετε οποιασδήποτε προτάσεις να μου κάνετε για να βελτιώσουμε το πώς θα ζούμε καλύτερα στην, στην περιοχή μας, στις πατρίδες μας, βοηθήστε με. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζον Καρλό Σκοτάλη, ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι έκλεισε το σημείο. Περιμένουμε τις τροπολογίες και στην επόμενη συνεδρίαση, 1η Δεκεμβρίου, θα υιοθετήσουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Τώρα, πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Είναι ένας ειδικός διαγνωστικός έλεγχος της Γεωργίας. Ο κύριος Ντόρφμα θα κάνει μια πρώτη παρουσίαση και συνεχεία θα ακολουθήσει μια συζήτηση για να συντάξουμε αυτή την ε, έκθεση πρωτοβουλίας που λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία. Όχι μόνο αυτό που το ελεγκτικό συνέδριο ε, μας είχε ζητήσει να κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική της έκθεση. Ε, και οι ορεινές περιοχές ανήκουν και εντάσσονται στο, στο πλαίσιο αυτής της ε, ειδική έκθεσης. Α, ένας εμπειρογνώμονας θα κάνει την παρουσίαση, ο κ. Ζόναρ, γιατί δούλεψε μαζί με τον εισηγητή η κυρία Ζώνα. Allora? Είναι ή δεν είναι η κυρία Ζώνα. ζωνα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας ζητήσατε να κάνουμε μια παρουσίαση για την ανακοίνωση του, α, της αναθεώρησης του καθεστώτος προς τις μειονεκτούσες περιοχές. Ε, συνεργαζόμαστε με τον εισηγητή του Κοινοβουλίου, αλλά εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι κάνετε λάθος στην παρουσίασή μου. Ε, θα ήθελα να σας εξηγήσω τα βασικά σημεία αυτής της ανακοίνωσης, η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο θα κάνω μια παρουσίαση ε, σε δύο τμήματα. Ένα πρώτο τμήμα είναι μια γενική παρουσίαση, γιατί κάνουμε αυτή την αναθεώρηση και σε τι σημείο βρισκόμαστε. Και σε, ένα δεύτερο, σε μια δεύτερη φάση θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση των ε, βασικών στοιχείων, δηλαδή νέα κριτήρια για τη ζωνοποίηση που μελετάμε και πώς θα καταστήσουμε την ε, βοήθεια πιο αποτελεσματική. Λοιπόν, έχω μία παρουσίαση PowerPoint, η οποία έχει προβλεφθεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να παρουσιάσουμε, αν έχουμε τις οθόνες για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση PowerPoint. Αν έχετε λάβει ε, επί χάρτου αυτή την παρουσίαση, θα δείτε ε, στο, στη δεύτερη διαφάνεια ένα χάρτη με τις μειονεκτούσες περιοχές, όπως τις προσδιορίζουμε αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε, η βοήθεια στου γεωργού σε αυτές τι μειονεκτούσε περιοχές είναι ένα κλασικό εργαλείο της ε, πολιτική ε, πολιτικής και ανάπτυξης ε, υπαίθρου ε, που ισχύει από το 1975 και είναι ένα καθεστώς που εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη παρά ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Και σε αυτή τη φάση ασχολούμαστε με, ένα, με μία μόνο από τις τρεις ε, μειονεκτούσες περιοχές. Δηλαδή, οι ενδιάμεσες ε, και ορεινές ε, ζώνες, περιοχές που έχουν ειδικά μειονεκτήματα, αυτές δεν τις ε, εντάσσουμε στην αναθεώρηση. Τώρα, οι ενδιάμεσες ζώνες, οι μειονεκτούσες που, σε οποίες εστιάζουμε υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από τη Δανία, τη Μάλτα και τις κάτω χώρες. Και λαμβάνουν για, μια περί... για την περίοδο προγραμματισμού που είναι εξελίξη, δηλαδή 2007-2013, ε, μια δημόσια βοήθεια που ξεπερνάει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 7,6% όλου των δημόσιων δαπανών που πηγαίνουν για την ανάπτυξη της υπαίθρου για αυτή την περίοδο προγραμματισμού. Ε, και είναι ε, αντισταθμιστικές αποζημιώσεις για αυτές τις μειονεκτούσες ε, περιοχές που δεν είναι όμως ορεινές. Είναι αυτές οι ζώνες σε κίτρινο σε αυτό το χάρτη και που είναι περίπου το 31% της γεωργικής επιφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών. Και οι εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν βοήθεια σε αυτές τις περιοχές είναι περίπου το 7% του συνόλου των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, θα περάσω στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια. Η αναθεώρηση που γίνεται αυτή τη στιγμή έχει πολύ συγκεκριμένη οριοθέτηση. Δεν πρόκειται να προτείνουμε μια νέα πολιτική, αλλά να αναπτύξουμε ένα πολιτικό εργαλείο το οποίο υπάρχει ήδη και είναι μια προσπάθεια ε, να επικεντρωθούμε στον ορισμό των ε, επιλέξιμων περιοχών και πώς θα προσανατολίσουμε καλύτερα τις βοήθειες αυτές, τη βοήθεια αυτή για να τις την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική. Αλλά δεν ασχολούμαστε με τις ορεινές περιοχές, το ξαναλέω. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη φάση προγραμματισμού δεν είναι ούτε να μειώσουμε, αλλά ούτε να αυξήσουμε τις τις, ορεινε, τις ε, μειονεκτούσες περιοχές. Απλώς την ταξινόμηση που κάνουμε ούτως ή άλλως θέλουμε να την κάνουμε πιο αντικειμενική και πιο διαφανή. Τώρα, για να καταλάβετε τη λογική αυτής της προσπάθειας, θα πρέπει να εξετάσουμε την εξέλιξη των στόχων αυτού του καθεστώτος βοήθειας προς τις μειονεκτούσες περιοχές. Είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει αλλάξει μέσα στη διάρκεια του χρόνου, όπως και η υπόλοιπη ΚΑΠ, για να προσαρμοστεί στις ε, αλλαγές της κοινωνίας. Το καθεστώς που δημιουργήθηκε το 1975 και αυτό που υπήρχε τον 20ο αιώνα είχε σαν σκοπό να διατηρήσουμε το φυσικό τοπίο και να αποφύγουμε την ε, απερίμωση των γεωργικών περιοχών. Σήμερα οι κοινωνικο-οικονομικοί στόχοι δεν ε, μπαίνουν έντονα στη λογική του καθεστώτος στη λογική αυτή της βοήθειας. Ε, θέλουμε απλώς να κρατήσουμε το φυσικό τοπίο για να συνεισφέρουμε σε μια βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και μια καλή διαχείριση γενικά του φυσικού τοπίου. Αυτή είναι μια εξέλιξη που θα πρέπει να τη δούμε υπό την ε, αιγίδα της ε, μεταρρύθμισης της ΚΑΠ του 2003 και της εισαγωγής μιας στρατηγικής διάσταξης, διάστασης του 2006, όπου άλλαξε η λογική των βοηθειών και εστιάστηκε στον δεύτερο άξονα, δηλαδή ε, προώθηση του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου. Εστιάσουμε περισσότερο εκεί τώρα από οπουδήποτε αλλού. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την διάσταση αυτή την περιβαλλοντική για τη διαχείριση του εδάφους, η βοήθεια των μειονεκτουσών περιοχών δεν είναι, δεν υπόκειται στα αγροεπιστητικά στοιχεία. Ε, αποφεύγει την απερίμωση των εδαφών ε, και όπου είναι δύσκολη η άσκηση της γεωργίας και τα αυταόχρονα αντισταθμίζει μόνο αυτό το μειονέκτημα και δεν καλύπτει το κόστος τον, το περιβαλλοντικό που έχει η γεωργία. Δηλαδή έχει μία ενδιάμεση θέση και διαφορετική σε σχέση με την ενιαία πληρωμή από τη μία και από την άλλη με τα μέτρα τα γεωργοπεριβαλλοντικά. Τώρα, για ποιο λόγο αυτή η αναθεώρηση ε, γίνεται τώρα. Το σημείο στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής σας μιλάει για ένα ειδικό διαγνωστικό έλεγχο. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες παθολογίες, κάποιες, κάποια προβληματικά σημεία ε, στο καθεστώς που υπάρχει και ότι σε γενικές γραμμές η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι στιγμή συμφωνούν ε, με τη διάγνωση αυτή ότι υπάρχουν αδυναμίες και είναι ένα καθεστώς το οποίο πρέπει να αλλάξει. Οι μειονεκτούσες ζώνες, οι ενδιάμεσα αυτές οι μειονεκτούσες περιοχές, ε, τα αξινομήθηκαν στο παρελθόν επί τη βάση Ενό συνόλου μιας δέσμη δικτών. Κάθε ένας από αυτούς τους δείχτε είναι κοινωνικονομικού χαρακτήρα, όπως παραδείγματο χάρη ε, η ένταση του πληθυσμού ή το μέσο εισόδημα. Και δεν συνάδουν πλέον με την σημερινή και σύγχρονη λογική α, του καθεστώτος. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη για να καθοριστούν αυτέ οι ζώνες είναι πάρα πολύ περίπλοκα και τελείω διαφορετικά μεταξύ του. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 100 κριτήρια ταξινόμησης των ε, περιοχών αυτών. Και επομένως υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας και ένας κίνδυνος ε, διαφορετικής μεταχείρισης. Κάτι που εντοπίστηκε και από το ελεκτικό συνέδριο. Παραδείγματος χάρη, η, ένταση, η μέγιστη ένταση του πληθυσμού, δηλαδή 15 15 κάτοικοι ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Εστονία, ενώ 130 στη Γερμανία. Με βάση την αξιολόγηση που έγινε πρόσφατα για το καθεστώς των ε, βοηθειών, λέμε, ε, προκύπτει ότι δεν πηγαίνει πάντα η πληρωμή σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται. Τώρα, σε τι φάση είμαστε με τη θεωρία, με την θεραπεία, συγγνώμη. Κάποια προβλήματα έχουν επιληθεί, αλλά το θέμα το που είναι δύσκολο, που είναι ο εντοπισμός και κυριοθέτηση των ε, περιοχών αυτών, αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ελεγκτικό συνέδριο μας ζήτησε να ξαναδούμε ε, άρδιν την ε, ταξινόμηση αυτών των ενδιάμεσων ε, ζωνών με βάση κοινά κριτήρια και το Συμβούλιο το 2005 ζήτησε από την Κομισιόν να κάνει μία ανάλυση και να κάνει προτάσεις. Η Κομισιόν, ακριβώς από αυτή τη βάση, δημιούργησε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων και αυτή η ομάδα μίλησε για 8 δυνατά κριτήρια κλιματικά νομίζω για να ταξινομήσουμε αυτές τις ε, περιοχές. Πρόκειται για κριτήρια που αφορούν το κλίμα, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, την κλίση και την ε, σχέση κλίματος και εδάφους. Είναι κριτήρια τα οποία αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία της ανακοίνωσης και θα τα βρείτε και στο τέλος του κειμένου που σας μοιράσαμε. Με βάση αυτή την τεχνική δουλειά που έγινε, έγινε μετά μία διαβούλευση μεταξύ κομισιών κρατών μελών και όλων των διαφερομένων μερών. Έγινε και μία δημόσια διαβούλευση το 2007 και εκατοντάδες συναντήσεις. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, τώρα είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τη βάσης, τις βάσεις δεδομένων που έχουν για να προσμετρήσουν την επίπτωση μιας νέας οριοθέτησης με βάση τα νέα κριτήρια. Γιατί η οριοθέτηση είναι κάτι το πολύ δύσκολο και ευαίσθητο. Και τα δεδομένα που έχουμε σε επίπεδο Κομισιόν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκό δεν, έχουν δεν έχουν το επαρκές επίπεδο λεπτομεριών. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν ασχοληθεί με την διαβίβαση χαρτών ε, με αυτές τις προσωμιώσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτή τη φάση ε, συνεργαζόμαστε με εθνικούς εμπειρογνώμονες για να δούμε αν όλες οι προσωμιώσεις αυτές μπορούν να είναι έτοιμες τον Ιανουάριο ούτω ώστε να μπορέσει η Κομισιόν να ολοκληρώσει μια ανάλυση επιπτώσεων και να εκπονήσει τελικά την πρότασή της. Τώρα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, με τα δεδομένα που έχουμε και με τη μέχρι τούδη ανάλυση που έχουμε κάνει, τα πλεονεκτήματα που βλέπουμε με αυτό το σύστημα που θα βασίζεται σε αυτά τα κοινά οκτώ κριτήρια είναι τα κάτω. Καταρχά, είναι ξεκάθαρο το σύστημα ε, που βασίζεται σε επιστημονικά διαφανή κριτήρια, ε, διαφανή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να καλύψει και τα φυσικά μειονεκτήματα που υπάρχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να απλουστεύσει τα πράγματα. Αρκεί μόνο ένα κριτήριο για να δούμε αν μια ζώνη είναι μειονεκτούσα. Ενώ μέχρι τώρα έχουμε πάνω από 100. Επίση όμω, οι εκατοντάδε συνεδριάσει που κάναμε με τα κράτη-μέλη μα επιβεβαίωσαν ότι ούτω ή άλλω τα κριτήρια είναι κατάλληλα και αξίζει να τα λάβουμε υπόψη. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι προσωμιώσει που θα κάνουν τα κράτη-μέλη για να κάνουμε την ανάλυση επιπτώσεων με πολύ ενδελεχή τρόπο. Τώρα, πέρα από τα 8 κριτήρια, τα κλιματικά, υπάρχει ένα στοιχείο που αναφέρεται στην ανακοίνωση και που αφορά την ανάγκη να εστιάσουμε τη βοήθεια. Δηλαδή, να τελειοποιήσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις την οριοθέτηση αυτών των μειονεκτουσών περιοχών. Σε ορισμένες περιοχές η επιστημονική ε, πρόοδος ή η ανθρώπινη παρέμβαση ε, βοήθησε ώστε να ξεπεραστούν τα, μειονεκτή, τα μειονεκτήματα, να έχουμε μια πολύ αποδοτική γεωργία. Έχω ετοιμάσει κάποιες φωτογραφίες με παραδείγματα, όπου παραδείγματο χάρη σε μια πολύ άγονη περιοχή, με την άρτευση μπορούμε να έχουμε μια γεωργία πραγματικά πολύ εντατική. Και οι επιπτώσεις ε, στο περιβάλλον βεβαίως μπορούν να συζητηθούν εδώ. Τώρα, σε ζώνες αντίθετα με προβλήματα υπερβολικού νερού, και με προσπάθειες παρέμβασης για να ε, διώξουμε τα νερά, μπορούμε να έχουμε επίσης μία επικερδή γεωργία. Συχνά έχουμε ε, ζώνες, ε, περιοχές ας πούμε, όπου έχουμε πάρα πολλές πέτρες και που με, μεγάλη προσπάθεια επί δεκαετίες καταφέρουμε να έχουμε προϊόντα πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το χάρτη των μειονεκτουσών ζωνών ε, δεν πρέπει να βάζουμε τις ζώνες που η γεωργία είναι πολύ επικερδής και μόνο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο το σύστημα δεν είναι αξιόπιστο. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο όχι για όλες τις περιοχές, αλλά για κάποιες περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα είναι απαραίτητο να τελειοποιήσουμε την οριοθέτηση των ε, περιοχών αυτών. Σε μια επόμενη φάση της ε, οριοθέτησης, αφού ο χάρτης των ε, περιοχών αυτών έχει ολοκληρωθεί, σε μια επόμενη φάση λοιπόν μπορούμε να εστιάσουμε την βοήθεια, να κάνουμε μια επιλογή δηλαδή των δικαιούχων και να δώσουμε τη βοήθεια μόνο στις εκμεταλλεύσεις που πραγματικά ε, κινδυνεύουν και μπορεί να καταληφθούν ε, και που βοηθούν στην ε, βιώσιμη διαχείριση των περιοχών. Αυτό δεν είναι καινοτομία. Το κάνουν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Ε, Όπω σα είπα, στι ενδεχτέ περιοχέ μόνο το 7% των γεωργών λαμβάνει βοήθεια. Αλλά δεν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο. Αυτό λείπει σήμερα για τα κριτήρια επιλεξιμότητα των και γι' αυτό λοιπόν διερωτώμεθα μήπως θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτό το κοινοτικό πλαίσιο για να υπάρξει καλύτερη εστίαση και να δούμε σε ποιον θα πάνε οι βοήθειες, ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι όχι. Θα τελειώσω με τις επόμενες φάσεις. Περιμένουμε τέλος του 2010 τις προσωμιώσεις των κρατών μελών Και αν η επόμενη Επιτροπή επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα, τότε θα υπάρξει μια πρόταση για τα νέα κριτήρια την επόμενη χρονιά, στο τέλος του 2010. Ρεαλιστικά, η νέα οριοθέτηση αποκλείεται να εφαρμοστεί πριν από το 2014. Θα τεθεί σε ισχύ λοιπόν αυτή η νέα οριοθέτηση ταυτόχρονα με τη θέση σε ισχύ του νέου συστήματος. Φυσικά, αν κάποιες περιοχές χάσουν το καθεστώ τους ως μειονεκτούσες περιοχές, αυτό δεν θα το ξέρουμε παρά μόνο όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι θα συμβεί σίγουρα. Και τότε μπορούμε να δούμε μήπως θα γίνει αυτό βαθμιαία ε, μήπως δηλαδή ο αποχαρακτηρισμός τους ε, μπορεί να γίνει βαθμία, να γίνει ένα phasing out. Ευχαριστώ την κυρία Τζόνα. Ζητώ συγγνώμη για το μπέρδεμα με το όνομα, Τζόνα, Τζόνα. Ε, νομίζω ότι είναι σαφές πλέον το πλαίσιο και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντόρφμαν και συνεχεία θα ακολουθεί η συζήτηση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, c'è da aggiungere poco, ringrazio la dottoressa Nazzona anche per la collaborazione nelle ultime settimane in quanto... Πολύ ωραία. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, δουλέψαμε πολύ για να παρουσιάσουμε αυτή την ε, έκθεση. Θα ήθελα να συνοψίσω πολύ σύ, σύντομα. Ε, Μιλάμε για τα κριτήρια της οριοθέτησης των μειονεκτουσών περιοχών. Ε, θα βασιζόμαστε όχι μόνο στα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια όπως γίνεται σήμερα, αλλά σε κριτήρια καθαρά κλιματικά. Σίγουρα υπάρχει μια ανάγκη ε, να ετοιμαστούν αυτές οι προσωμιώσεις που τις περιμένουμε τέλος Ιανουαρίου από, την Ευρωπαϊκή, από τα κράτη-μέλη, τα περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα στοιχεία και θα δούμε μόνο τι επίπτωση θα έχουν αυτά τα κριτήρια, τα οποία είναι πολύ επιστημονικά. Αλλά μόνο αφού έχουμε τις ε, προσωμιώσεις θα είμαστε σίγουροι. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Και συνεχεία στη συζήτηση θα προκύψουν σίγουρα και άλλα στοιχεία. Φυσικά, θα πρέπει να συζητήσουμε αν αυτά τα 8 κριτήρια είναι σωστά, αν είναι επαρκή για να κάνουμε με δίκαιο τρόπο αυτή την ε, οριοθέτηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, είναι σωστές οι μέθοδοι μέτρησης. Η πρόταση της Επιτροπής ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα κριτήριο, ας πούμε, θα πρέπει να είναι πραγματικότητα τουλάχιστον στα δύο τρίτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα 2 τρίτα, αυτό το 66% είναι πολύ υψηλό νούμερο, πολύ χαμηλό νούμερο. Δεν ξέρουμε. Επίσης, πρέπει να αξιολογήσουμε ε, κάποια σορευτικά στοιχεία. Δηλαδή, αν έχουμε δύο και 3 ή και περισσότερα κριτήρια μειονεκτήματος. Αφρίζουμε λοιπόν έτσι διάφορα μειονεκτήματα. Ε, πρέπει να το κάνουμε όμως αυτό, να κάνουμε αυτό τη συσσόρευση ή όχι. Προς το παρόν η Κομισιόν δεν προβλέπει αυτή την, αυτό το στοιχείο της συσσόρευσης. Η κυρία Τζόνα μας είπε ότι για το κριτήριο το κλιματικό και του εδάφους. Για σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη τις αμπελουργικές ε, περιοχές ή τις περιοχές με ελιές. Συχνά όμως το φτωχό, το φτωχό έδαφος ας πούμε δημιουργεί καλύτερη παραγωγή. Ε, θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να χτενίσουμε τα κριτήρια αυτά σε επίπεδο κρατών μελών, ούτω ώστε να αποκλείσουμε αυτές τις πολύ επικερδείς περιοχές από την οριοθέτηση που κάνουμε. Επίσης, το θέμα του phasing out. Μια και μιλάμε για νέα, νέο προσδιορισμό των περιοχών. Ε, προφανώς κάποιες θα μπουν σε αυτή τη νέα οριοθέτηση και κάποιες θα βγουνε. Για αυτές που βγαίνουν, θα πρέπει να γίνει ε, αυτή η αποχώρηση, αυτό, αυτή η διαγραφή τους ε, βαθμιαία. Πόσο θα διατηρηθεί, σε τι, πώς θα γίνει αυτό το phasing out, πόσο περιοδικ, προοδευτικά συγγνώμη, και βαθμιαία θα, θα βγούνε από τις σημερινές ε, περιοχές. Έπειτα, για το χρονοδιάγραμμα. Ε, αυτή η έκθεση θα ολοκληρωθεί είτε το Δεκέμβριο είτε τον Ιανουάριο. Δηλαδή θα, θα τελειώσουμε πολύ γρήγορα, είναι στενό το χρονοδιάγραμμα, επομένως συνεργαστείτε παρακαλώ για να είμαστε παραγωγικοί. Η κυρία Γκαρσία Πέρες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Ντόρφμαν για την παρουσίαση που μας έκαναν αυτή της πρότασης για τις μειονεκτικές περιοχές. Θα είμαι ιδιαίτερα λακωνική. Θα ήθελα απλώς να σας διαβιβάσω μία ανησυχία που προέκυψε από τις αλλαγές ε, της ανακοίνωσης ευρωπαϊκής περιοχής. Γιατί ε, διαγράφοντας τα κοινωνικο-οικονομικά κριτηρία αποκλεί ουσιαστικά τις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού για, πολλές, για πολλούς φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία από τις μείζονες προκλήσεις αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απερίμωση και ιδιαίτερα η εγκατάλειψη ορισμένων ε, γεωργικών περιοχών και η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ε, γι' αυτό διαγράφοντας το, κριτήριο του αεροκατοικημένου, της αεροκατοικημένης ζώνης, της χαμηλής πυκνότητας, μήπως ε, αυξήσουμε το μειονέκτημα αυτών των περιοχών που όλο και λιγότερα όλο και λιγότερες δυνατότητες δίνουν στην νεολαία τους για να, παραμείνουν, για να παραμείνει στην περιοχή αυτή. Από το χάρτη που μας προτείνατε θα δούμε πώς έχει κατάσταση στα κράτη-μέλη και ποια θα είναι η επίπτωση των αλλαγών που προτείνεται στην ανακοίνωση για τις μειονεκτικές περιοχές. Θα δούμε και από τις προτάσεις των κρατών μελών τι το οποίο θα δημιουργηθεί για να λάβουμε και εμείς θέση. Πάντως, αν μία από τις προκλήσεις αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός στην ύπεθρο που καθημερινά ε, φιλορροεί και χάνει τους νέους της που μετακινούνται προς ε, μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Αν αφαιρώντα ε, το κριτήριο της χαμηλής του πληθυσμού, στερούμε και αυτή τη δυνατότητα από τις περιοχέ, νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με την ανακοίνωση. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή, γιατί πρέπει να γίνει ένας διαγνωστικός έλεγχος στις ζώνες με φυσικά μειονεκτήματα. Έχουμε επίγνωση της δυσκολίας που έχει δημιουργία κάποιων κριτηρίων ταξινόμησης που θα είναι ικανοποιητικά για όλους. Πάντως, συμμεριζόμαστε ένα κοινό στόχο, να αποφευθεί απερίμωση, εγκατάλειψη των περιοχών και ιδίω από τους νέους. Αλλά υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Όταν μιλάμε για, τη βοήθεια αντιστάθμισης ε, ε, και των παράγωγων ε, προβλημάτων από τα φυσικά μειονεκτήματα. Έγινε σωστή καταμέτρηση των επιπτώσεων πέραν των κριτηρίων της διαφάνειας και της καλύτερης διαχείρισης που φυσικά συμμεριζόμαστε. Αυτές οι οριοθετήσεις έλαβαν υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχουν τα μέτρα αυτά στις ζώνες που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται ως ενδιάμεσες μειονεκτικές ε, περιοχές. Επίσης, ε, η κυρία Γκαρσία Πέρες είπε, αν αφαιρεθούν τα οικονομικοκοινωνικά κριτήρια και δεν ληφθούν υπόψη ε, οι ζώνες που δεν έχουν άλλες εναλλακτικές παραγωγής, αποκλείται να αποφύγουμε την εγκατάλειψη του πληθυσμού και θα επιτείνουμε δίνει η κατάσταση που δημιουργείται με τα φυσικά μειονεκτήματα. Τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια είναι αντικειμενικά κριτήρια. Γιατί να μην παραμείνουν και αυτά στο κατάλογο, αποκοινούμε τα υπόλοιπα κριτήρια που, που προτείνουν οι βιοφυσικοί. Τα βιοφυσικά κριτήρια δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι υψηλό ή χαμηλό το ποσό των το 66% ε, ως προς την ε, ωφέλιμη γεωγραφική έκταση. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικό αυτό το κριτήριο του 66%. Και κάτι άλλο που με προβληματίζει και με ανησυχεί τα μάλα είναι η πρόταση να αποκλειστεί από τον κατάλογο αυτό των ενδιάμεσων μειονεκτικών περιοχών οι περιοχές που με την παραγωγή και τα τεχνικά μέσα ξεπέρασαν τα φυσικά τους μειονεκτήματα. Μα αυτό δεν έχει νόημα. Αυτός που κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να ξεπεράσει τα φυσικά διαρθρωτικά μειονεκτήματα που έχει, που όμως δεν τα έχει αποκλείσει. Μπορεί να κατάφερε να τα ξεπεράσει μια δεδομένη στιγμή αυτά τα φυσικά μειονεκτήματα, αλλά δεν τα έχει εξαφανίσει. Άλλωστε το κόστος είναι τεράστιο. Γιατί να τις τιμωρήσουμε λοιπόν αυτές τις περιοχές που έκαναν τέτοιες κολοσσιαίες προσπάθειες για να ξεπεράσουν το φυσικό τους μειονέκτημα αντί να τις επιβραβεύουμε, να τις ε, τιμωρούμε αφαιρώντας τις από το κατάλογο, γιατί τους θερούμε τα δικαιώματα ενίσχυσης για, για τα μειονεκτήματα που είχαν. Έχουν ε, εξοβελιστεί και οι ορεινές περιοχές ε, και άλλες με ιδιαιτερότητες εγώ πιστεύω ότι και οι ορεινέ περιοχές και οι υπεραπόκεντρε περιοχές βέβαια χρήζουν ιδιαίτερη μεταχείρισης σε ορισμένε περιπτώσεις, αλλά γιατί να αποκλείονται ρητά από τον χαρακτηρισμό των ενδιάμεσων μειονεκτικών περιοχών. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα αυτών των ζωνών είναι πολύ σημαντικά, πέραν του σοβαρού προβλήματος που έχουμε με το νερό και μάλιστα πολύ συχνά επιδεινώνονται αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Γι' αυτό και τα μειονεκτήματά τους είναι σημαντικά. Γιατί λοιπόν να αποκλειστούν από τις ενδιάμεσες μειονεκτικές περιοχές. Ευχαριστώ κύριος Άλμπερτ Ντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο που έθιξε αυτό το που επεξεργάστηκε το θέμα αυτό και θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η συζήτηση πρωτού καταλήξουμε σε μια σωστή λύση. Να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να είναι εντατική η συνεργασία μας προκειμένου να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα είναι κοινά αποδεκτή. Για παράδειγμα, εμείς από τις ορεινές περιοχές έχουμε όλα τα υψόμετρα ουσιαστικά στην Βαυαρία, σχεδόν και να σας πω ότι ως τώρα ενίσχυση των μειονεκτούσεων περιοχών ήταν με πολύ ε, ανεπιτυχής, με πολύ πιο μικρά, με πολύ πιο περιορισμένα μέσα, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα σωστό σύστημα. Δεν μπορούμε να παράγουμε ένα σύστημα γραφειοκρατικό, μόνο και μόνο για να προάγουμε τις ε, περιοχές με μειονεκτήματα. Θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα, ένα σύστημα με 100 σημεία για παράδειγμα, που θα μπουν τα κριτήρια Όποια περιοχή έχει για παράδειγμα πληρεί 100 κριτήρια θα έχει το 100%. Όποια περιοχή έχει 20 κριτήρια το 20% και το καθεξής και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα αποβεί προς το συμφέρον όλων μας. Δηλαδή, με τα ευρωπαϊκά μέσα και τη συγχρηματοδότηση να εξεύρουμε το σύστημα εκείνο με το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα τους γεωργούς στις ε, μειονεκτικές αυτές περιοχές προκειμένου να τονίσουμε, να τονώσουμε και τον ανταγωνισμό και να μπορέσουμε με καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτούμε στο μέλλον τις περιοχές αυτές. Albert. Ευχαριστούμε, Albert. Ο κύριος Σμιθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ε, ζητώντας συγγνώμη που άργησα. Δεν παραβρέθηκα εδώ στην αρχή της συζήτησης, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να βρίσκομαι σε δύο σημεία και μπήκα στα μέσα της παρουσίασης της Επιτροπής. Ωστόσο, το θέμα αυτό το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, ιδιαίτερα επειδή είμαι από τη Σκοτία όπου έχουμε νησιά με χαμηλή πυκνότητα και με μεγάλη οικονομική δράση. Προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ τα θέματα αυτά και από ό,τι φαίνεται και ο εισηγητής ε, προσέχει το θέμα αυτό. Θα συμφωνήσω με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για την αφαίρεση των κοινωνικών κριτηρίων στη μεταρρύθμιση του πακέτου αυτού, γιατί πρόκειται για ένα μηχανισμό κατεξοχή ε, κοινωνικό οικονομικό. Δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν αυτοί οι στόχοι και μιλάμε για την απερίμωση, μιλάμε για τη διατήρηση των κρίσιμων υποδομών σε θέματα παραγωγής σε περι, περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού και να, κοιτάμε ότι δεν μιλάμε, να κοιτάξουμε ότι δεν μιλάμε για ε, χοντρική μεταρρύθμιση του συστήματος, γιατί πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Το γεγονός ότι κοιτάμε τη μεταρρύθμιση του συστήματος LFA είναι ότι έχει γίνει κατάχρηση του συστήματος σε άλλα κράτη-μέλη. Γιατί το σύστημα LFA αποσκοπεί στην ενίσχυση περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και γι' αυτό πιστεύω ότι η εργασία αυτή που πρόκειται να κάνουμε έχει τη δυνατότητα να αποβεί προς όφελος των μειονεκτούντων περιοχών αυτών, γιατί αυτό είναι που μετράει για όλους μας, η διατηρήση της σε αυτές τις ε, περιοχές. Νομίζω ότι είναι κρίσιμη αυτή η στιγμή και καλό είναι που επανεξετάζουμε αυτό το θέμα. Σήμερα είναι προφανές ότι πολλές γεωρικές εκμεταλλεύσεις ε, θεωρούν τις ενισχύσεις ως συμπλήρωμα του εισοδήματός τους. Οπο, οποιοςδήποτε ε, αποχαρακτηρισμός ή αλλαγή του χαρακτηρισμού τροποποιεί και τον αριθμό των ε, δικαιούχων της ενίσχυσης. Ποιος ε, θα λάβει την απόφαση για τον αποχαρακτηρισμό μιας ζώνης και ποιος θα την εξηγήσει, γιατί όταν υπάρχει κρίση στην παραγωγή θα πρέπει να είμαστε λογικοί στην υποστήριξη των επιχειρημάτων και στον και των Έχω και κάτι άλλο υπόψη που δεν έχει συμπεριληφθεί στη, στην προσπάθεια αυτή. Πρόκειται για ζώνες που εξαιτία της εντατικοποίησης ε, ε, ή εξαιτία της λειψιδρίας ε, βρέθηκαν σε καταστάσεις ολέθριες. Γιατί εξαιτία υπερβολικής άρδευσης εξαντλήθηκε ο υδάτινος ορίζοντας, ε, για παράδειγμα για την παραγωγή αραβόσιτου. Και εξαιτία αυτής της ε, ε, υπερβολικής και εντατικής γεωργίας, οι ζώνες αυτές βρέθηκαν σε πολύ ευπαθή κατάσταση και πρέπει να συνταχθούν. Χρησιμοποιήθηκαν κάποιες γεωργικές πρακτικές που αυτό σε φτώχηση το εδάφους. Θα πρέπει να εφαρμόζουμε γεωργικές πρακτικές που θα σέβονται το έδαφος πέραν των κλιματικών συνθήκων. Χρειαζόμαστε κάποιες γεωργικές περιοχές, ε, γεωργικούς τρόπους παραγωγής που θα σέβονται το έδαφος και το περιβάλλον. Και κλείνει παρεμβάσεις με τον, με τον τελευταίο μιλητή Καπούλα Σάντος. Μάλλον δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει μια ευρυθή συζήτηση. Πάντως το θέμα που εξετάζουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα μοντέλο με δύο είδη ε, ενισχύσεων. Το, σύστημα, το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ευνοεί τις περιοχές που έχουν περισσότερα θετικά στοιχεία και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη κάποια ιστορικά κριτήρια που ενισχύει αυτές τις περιοχές ακόμη περισσότερο. Ενώ το καθεστώς ενισχύσεων για, για τα φυσικά μειονεκτήματα προσπαθεί να ευνοήσει περιοχές που είναι μειονεκτικές. Η συζήτησή μας λοιπόν θα πρέπει να είναι ακόμη πιο φιλόδοξη. Γιατί βρισκόμαστε στις παραμονές της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Αυτό το, νέο γεωργικό κοινοτικό μοντέλο θα πρέπει να καλύπτει όλα αυτά τα συστήματα των ενισχύσεων δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε σε ένα σκέλος μόνο, ούτε να διονίζουμε το παλιό μας μοντέλο. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι απαραίτητο να αλλάξουν όλα και να παραμείνουν όλα όπως έχουν. Δεν θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή τη λογική. Πολύ ωραία αυτά τα στοιχεία που προτείνετε για την συζήτηση, αλλά θα πρέπει να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε για να διαμορφώσουμε το νέο γεωργικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ίσως θα πρέπει να στηρίζεται σε έναν ενιαίο πυλώνα και θα έχει ένα σαφή κατάλογο κριτηρίων για τις ενισχύσεις, είτε για τις παραγωγικές ζώνες, είτε για τις μειονεκτικές περιοχές. Είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για την ε, εκτενή συζήτηση που θα πρέπει να διεξαχθεί και που θα πρέπει να είναι πολύ πιο σφαιρική, πολύ πιο ευρεία για ένα νέο γεωρικό μοντέλο. Δεν αρκεί να εμβαθύνουμε σε ορισμένα μόνο σημεία και να αλλάζουμε περιπτωσιολογικά το γνωστό μας μοντέλο. Θέλουμε άρδιν αλλαγή του γεωρικού μας μοντέλου. Ευχαριστώ πάντως τον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβολή του σε αυτή τη συζήτηση που πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο διευρυμένη γιατί με τη νέα νομική κατάσταση θα έχουμε και πολύ πιο ενισχυμένες εξουσίες. Στο Λουίς, ο εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Χόφμαν, ζητάει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω εν συντομία να απαντήσω στα ερωτήματα που μας θέσατε. Καταρχάς, θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι επειδή η διαδικασία αυτή επεξεργάζεται μόνο τις ενδιάμεσες μειονεκτούσες περιοχές, δηλαδή όχι τις ορεινές και όχι τις ε, ε, μειονεκτούσες περιοχές με συγκεκριμένα μειονεκτήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται η υποστήριξη για τις περιοχές αυτές, τις δύο τελευταίες αυτές περιοχές η διαδικασία αναθεώρησης χρησιμοποιείται μόνο σε αυτές τις ενδιάμεσες ζώνες ιδιαιτέρως, επειδή θεωρούμε και το επιβεβαιώνουν και άλλες αποφάσεις, όπως αποφάσεις και του ελεκτικού συνεδρίου, σε ό,τι αφορά τις ορεινές περιοχές και τις περιοχές με συγκεκριμένα μειονεκτήματα, όπως τα νησιά για παράδειγμα, δεν υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τον ορισμό και την διάκριση των περιοχών αυτών. Υπάρχουν πιο σαφή κριτήρια και δεν υπάρχουν ε, προβλήματα. Άρα δεν τα συζητάμε, δεν συζητάμε τις περιοχές αυτές. Σωστά ορίζονται, θεωρούμε, ως προς τα αντικειμενικά στοιχεία οι ορεινές περιοχές. Συζητάμε λοιπόν μόνο τις ε, ενδιάμεσες αυτές μειονεκτούσες περιοχές. Το δεύτερο στοιχείο για τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των ε, περιοχών αυτών αποτελεί μία από τις βασικές ανησυχίες της ε, πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Όπως ξέρετε, στις πολιτική υπάρχει ένα πλαίσιο πολιτικής ε, ανάπτυξης της υπαίθρου, το οποίο περιλαμβάνει 40 περίπου μέτρα, το οποίο, πολλά εκ των οποίων εστιάζονται στα κοινωνικο-οικονομικά μέτρα αλλά θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι τα μέτρα με τα οποία μπορούμε να καταπολεμήσουμε την απερίμωση, την εγκατάλειψη της υπαίθρου των περιοχών αυτών. Θεωρούμε ότι η ενίσχυση προς τους αγρότες για να διατηρήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους σε ευπαθείς περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα είναι κάτι διαφορετικό και το βασικό είναι να διτηρηθεί η καλλιέργεια, η εκμετάλλευση στην Ήπεθρο, στην περιοχή αυτή και πληρώνουμε το επιπλέον κόστος στον αγρότη. Αλλά η διατήρηση της αγροτικής εκμετάλλευσης, από ό,τι ξέρετε, δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των περιοχών αυτών. Υπάρχουν και άλλα απαραίτητα στοιχεία, όπως η απασχόληση, οι υποδομές όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερα για τους νέους, για τους πρεσβύτερους, προκειμένου να μένουν στις περιοχές αυτές, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια ποιότητα ζωής, να μην εξαναγκάζονται να προσφεύγουν στις πόλεις. Θεωρούμε ότι το μέσο αυτό για τις ε, λιγότερο ευνοημένες ε, περιοχές θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το στόχο του, την ενίσχυση δηλαδή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και σε ό,τι αφορά την ε, κατάσταση την κοινωνικο-οικονομική θα πρέπει να πάμε και να κοιτάξουμε πέρα από το μέσο αυτό, να δημιουργήσουμε άλλα μέτρα, άλλα μέσα για την απασχόληση, για τη βελτίωση της κατάστασης ε, στον κλάδο των τροφίμων, και για όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται για να διατηρηθούν βιώσιμες οι περιοχές αυτές. Από ό,τι είδατε, το εγχείρημα είναι αρκετά τεχνικής φύσεως, γι' αυτό συγχωρέστε με αν κάποιες φορές είναι δύσκολο να συγκεντρώσουμε όλα τα τεχνικά στοιχεία επί του θέματος, αλλά ένας στόχος μας ήταν σε τελική ανάλυση να καταλήξουμε σε ένα απλό σύστημα. Ένα σύστημα που δεν θα είναι περίπλοκο. Ασφαλώς και είδατε ότι στην πραγματικότητα χρειάζονται κάποιο, κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες διακρίσεις, ε, την ανάπτυξη κάποιων δικτών για τον ε, καθορισμό των περιοχών. Θεωρούμε ότι το σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο βάσει των οκτώ ε, αυτών κριτηρίων αποτελεί μια καλή βάση, αλλά θα πρέπει να εξαιρεθούν περιοχές, για παράδειγμα, όπου συστηματικά η πλειοψηφία των αγροτών δεν αντιμετωπίζει τα μειονεκτήματα αυτά, γιατί για παράδειγμα υπάρχει αποστράγγιση ή γιατί θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ενισχυθούν αυτοί οι αγρότες, να επικεντρωθούν τα κονδύλια σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες, όπου πραγματικά δυσκολεύονται οι αγρότες να συνεχίσουν την εκμετάλλευσή τους, γιατί δεν μπορούν να ανατρέψουν αυτό το μειονέκτημα, ούτε μπορούν να εγκαθιδρύσουν μια παραγωγή εξίσου ευνοϊκή όπως σε άλλες περιοχές. Στη συνέχεια, το θέμα της ε, σώρευσης των κριτηρίων. Να σχολιάσω το εξής. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει κανείς τρεις διαφορετικές δυσκολίες σε μια περιοχή και αν η πλειονότητα της περιοχής αντιμετωπίζει τις τρεις αυτές δυσκολίες, θεωρείται ως λιγότερο ευνοούμενη η περιοχή αυτή. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο δεν χρειάζεται ε, μία περιοχή να καλύπτει όλο το φάσμα των δυσκολιών. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι δείκτες. Δεν μπορεί να πούμε όμως, είναι δύσκολο να πούμε ότι αντιμετωπίζω ένα μειονέκτημα κατά 50%, κατά ένα άλλο κατά 20% και ένα τρίτο κατά 30% και όλα αυτά αντιστοιχούν σε 100%. Γιατί η υπεύθυνη κατάρτιση του συστήματος αναφέρουν ότι είτε φτάνει κανείς σε ένα επίπεδο μειονεκτήματος, είτε δεν αντιμετωπίζει μειονέκτημα. Αυτή είναι η αρχική θέση και φυσικά βρισκόμαστε σε φάση συζήτησης και με τα κράτη-μέλη και με εσάς, όπου θα πρέπει να εξετάσουμε φυσικά τα εκκρεμή ζητήματα για να διευκρινίσουμε την κατάσταση. Αλλά και για να αναπτυχθεί περαιτέρω το σύστημα το οποίο υφίσταται ήδη στα κράτη-μέλη. Ωραία, ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές, φυσικά και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι φαίνεται, πολύ πλούσια. Ε, γι' αυτό καλή τύχη και στον κύριο Ντόρφμαν για τη δουλειά του. Ε, κλείνουμε τώρα εμείς και εμείς θα τα ξαναπούμε στις 10. Στις 10